εν ώψη του ε, Συμβουλίου του ε, Δεκεμβρίου που θα ε, αφορά ακριβώς θέματα ασφάλειας. Πρόκειται για δύο εκθέσεις οι οποίες έχουν τη φιλοδοξία να εκπροσωπήσουν τη θέση του Κοινοβουλίου. Έστω και αν η γνώμη του Κοινοβουλίου δεν ζητάται απαραίτητα από τα κράτη-μέλη, εν πάση περιπτώσει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σε δύο λεπτά με αυτά τα θέματα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα όμως να σας ε, πω δύο λόγια όσον αφορά την αποστολή που κάναμε ε, σαν Επιτροπή, Υποεπιτροπή ΣΕΔΕ στη Γεωργία τον Ιούλιο. Η Άννα Γκόμες που είναι και εδώ σήμερα ήταν ε, μαζί μου, μαζί με τον Χριστό avec nous. Euh, oui, euh, Και είχαμε και την Τερέζα μαζί μας. Πρόκειται για μια αποστολή η οποία στόχο είχε όχι ακριβώς να αξιολογήσει την πολιτική κατάσταση στη Γεωργία βέβαια, έστω και αν πολλά θα μπορούσε να πει κανεί για το θέμα αυτό, αλλά ε, επικεντρώθηκε στην ε, αποστολή ε, επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2008 μετά από τη διένεξη μεταξύ Γεωργία και Ρωσίας. Στην ουσία λοιπόν συναντήσαμε τους εκπροσώπους αυτής της αποστολής επιτήρησης ε, καθώς επίσης και με εκπροσώπους της πολιτικής της Γεωργίας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε ε, να συναντήσουμε τον ε, Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας γιατί οι συναντήσεις αυτές την τελευταία στιγμή ακυρώθηκαν για λόγους απολύτως επισήμους όπως μας παρουσιάστηκαν αλλά που δεν μας έπεισαν παρόλα αυτά και που τελικά ε, δίνουν μια ιδέα της μεγάλης πολιτικής πόλωσης που διαπιστώσαμε επί τόπου και που είναι ιδιαίτερος ανησυχητική. Τον ε, προηγούμενο Οκτώβρη είχαμε χαιρετήσει αυτήν την ειρηνική ε, και μέσω αναμφισβήτητης της εκλογής του πρωθυπουργού στις τότε εκλογέ, αλλά δυστυχώ διαπιστώσαμε ότι το πολιτικό κλίμα στη Γεωργία δεν έχει αποκατασταθεί καθόλου μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει και οι συζητήσεις μας και οι επαφές μας δεν ε, έγιναν τελικά όπως είχαμε αρχικά ε, θεωρήσει. Παρ' όλα αυτά είχαμε την ευκαιρία να δούμε ότι η αποστολή επιτήρησης λειτουργεί επί τόπου ότι αξιολογείται θετικά η παρουσία αυτής της αποστολής και από πλευράς κυβερνήσεων ίσως και από πλευράς Προέδρου αλλά και πολιτικής αντιπολίτευσης γιατί όλοι υπογράμμισαν την σημασία αυτής της ε, αποστολής, αυτής της αντιπροσωπείας που είναι η μόνη ξένη διεθνής αποστολή η οποία διαθέτει την απαραίτητη νομιμότητα που της δίνει την δυνατότητα να δρά σε αυτό το ιδιαίτερα περίπλοκο ε, και τεταμένο περιβάλλον της Γεωργίας, της Οσετίας και της Αμπχαζίας επί που είχαμε ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις με πολλές ομάδες αυτές της αποστολής ε, διαπιστώσαμε από μόνοι μας αυτήν την διαδικασία η οποία ονομάζεται συνοριοποίηση ε, και ε, που ε, οι συνοριοφύλακες οι Ρώσοι και οι ε, ομάδες του στρατού ε, της Ρωσίας προσπαθούν σιγά σιγά να τρώνε ας πούμε λίγο από το έδαφος και να το περιφράσουν με φράγματα και με συστήματα επιτήρησης κτλ. Πάντως ε, διαπιστώσαμε ότι όλοι όσοι εργάζονται στην αποστολή ε, είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ε, όσον αφορά το ίδιο το προσωπικό και το δυναμικό μάλλον, εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Αυτή τη στιγμή είναι εκεί 300 άτομα αναρωτιέμαι εάν ε, μια αποστολή τόσο μεγάλου μεγέθους ε, δικαιολογείται, ε, έχει επιμηκυνθεί, έχει παραταθεί η διάρκεια ζωής της αποστολής. Εν πάση περιπτώσει έχουμε εδώ και εκπροσώπους οι οποίοι τον κύριο Κλάρ και την άλλη κυρία που είναι εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ξαναδούμε βεβαίως στην ε, Επιτροπή μας. Ε, θα είστε επικεφαλής αποστολής, μιας αποστολής η οποία και είναι σημαντική και στηρίζεται και από τα κράτη-μέλη και από την χώρα αποδέκτη, ε, αλλά και από τους πιο απομακρυσμένους, ας το πούμε, παρατηρητές. Ε, είναι μια αποστολή η οποία διαμφισβήτητα έχει και χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό ήταν και το μήνυμα που θελήσαμε να ε, περάσουμε. Θα δείτε εσείς ε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε το ζήτημα του προσωπικού, του αριθμού του προσωπικού, ενδεχομένως να κάνετε μια εκ νέου αξιολόγηση έτσι ώστε να δείτε ποιο ακριβώς είναι το προσωπικό που χρειάζεται. Τώρα το πρόβλημα και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και προς τα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα και στην ύπατη εκπρόσωπο και στον ε, προεδρεύοντα του Συμβουλίου και στον πρόεδρο της Επιτροπής διαπιστώνουμε ότι στον διάλογο με την Ρωσία δεν υπάρχει υπάρχει, ο, δεν ε, ε, τηρείται ο απαραίτητος σεβασμός των αρχικών ε, συμφωνιών. Η δυνατότητα λοιπόν ε, πρόσβασης στα εδάφη της Οσετίας και της Απχαζίας αποτελούν πάντοτε παράβαση, ε, παραβίαση συγγνώμη, των συμφωνιών του 2008. Δεν είναι δυνατόν μία ε, αποστολή ευρωπαϊκή η οποία έχει συγκεκριμένο καθεστώς και η οποία έχει γίνει αποδεκτή βάση ε, συμφωνιών να μην έχει ε, την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε αυτά τα εδάφη. Εμείς έχουμε συναντήσει και τους αρμοδίους από τη ρωσική πλευρά και πριν από λίγο καιρό στο Εκατερίνα Μπουργκ αλλά φαίνεται ότι δεν αποτελεί αυτή η περιοχή σημαντική προτεραιότητα. όλα αυτά είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να ρίξει και το φως της δημοσιότητας ε, στον ε, Κάφκασο. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι ε, πρέπει διαρκώς να υπενθυμίζουμε στην ρωσική πλευρά ότι υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες δεν γίνονται σεβαστές. Οι συμφωνίες του 2008 σε κάθε περίπτωση πρέπει να το αναφέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει εγώ αμφιβάλλω και κατά πόσον τα πράγματα θα βελτιωθούν ε, και εγώ δεν θεωρώ ότι ε, πιέζουμε αρκετά. Άλλωστε διάβασα και τα πρακτικά της ε, εαρινής συνάντησης διάσκεψης κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Δεν έχω την αίσθηση ότι πιέζουμε αρκετά. Πάντως είναι ανησυχητική η κατάσταση στη Γεωργία ακόμα. Πέρα από την ίδια την αποστολή εμείς συναντήσαμε και τον ε, Μεραβισβίλη, τον πρώην ε, Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι φυλακισμένος. Ε, διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να δεχτεί οικογενειακές επισκέψεις. Αυτό αποτελεί βεβαίως παραβίαση των δικαιωμάτων του. Μέσω της δικής μας πίεσης και μεσολάβησης αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα πρόβλημα. Επίσης συναντήσαμε και την ε, Υπουργό Δικαιοσύνη ε, της ε, Γεωργίας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση. όλα αυτά νομίζω ότι το σύνολο της αντιπροσωπείας, όλοι οι εκπρόσωποι δηλαδή, των πολιτικών ομάδων διαπιστώνουν με ανησυχία ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διαφθορά οπωσδήποτε και όσον αφορά αυτή την ακραία πόλωση του πολιτικού <coughs> συστήματος που <coughs> είναι μια ε, ιδιαίτερα ανησυχή κατάσταση. Διαπιστώσαμε ε, επί τόπου ότι ε, η ίδια η αποστολή δεν ενοχλείται ας πούμε από αυτήν την κατάσταση είναι δύο ξέχωρες καταστάσεις αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα, ιδιαίτερα προσεκτικοί πρόκειται για μια εξαιρετικά εμβληματική αποστολή για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ξέρετε ε, υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι οι αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι είτε επιφανειακές είτε στην ουσία επικαλύπτουν ή επικαλύπτονται από άλλες αποστολές άλλων οργανισμών. Σε τούτη εδώ την αποστολή επιτήρησης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ούτε ο ΑΣΕ, ούτε η, οποιαδήποτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κάποιος άλλος φορέας δεν έχει μια τέτοια αποστολή η οποία να αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας και να είναι ε, και συμφωνημένη και ε, θεσμικά ε, καλυμμένη. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε όταν αναρωτιόμαστε ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιες περιπτώσεις ενδυνάμωσης της πολιτικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Άννα θέλει να πει κάτι, ήταν μαζί μας. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που μας έκανε ο Πρόεδρος και με τα σχόλια που ακούσαμε. Θα ήθελα απλώ να επισημάνω ότι για αυτή την αποστολή που είναι ιδιαίτερα σημαντική, χρήσιμη και αναγνωρισμένη σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική πόλωση που υπάρχει στη χώρα δεν επηρεάζει την γενική υποστήριξη αυτής της αποστολής. Βέβαια η υποστολή αυτή ε, είναι δυνατή, αλλά θα, ε, είναι απαραίτητη η στρατητική εμπειρία των μερών αυτής της αποστολής, παρόλο που είναι πολιτική. Και θυμάμαι μια πολιτική αποστολή που είχαμε πολύ σημαντική και αποφασιστική σημασία για την ειρηνευτική διαδικασία Και εκεί ήταν χρήσιμη η στρατιωτική πείρα κάποιων μελών της αποστολής. Γιατί φυσικά χρειάζονται και η εμπειρία σε μη στρατιωτικά θέματα, αλλά και η εμπειρία σε στρατιωτικά ζητήματα. Γιατί μερικοί που έχουν στρατιωτική πείρα βλέπουν πράγματα που οι υπόλοιποι δεν βλέπουν και γι' αυτό είναι πολύτιμη αυτή η πείρα. Και τα θετικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στρατιωτική πείρα κάποιων μελών της αποστολής. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είναι ανησυχητική αυτή η πολιτική πόλωση που διαπιστώνουμε στη Γεωργία. Και ήταν χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό της Γεωργίας. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το γενικό κλίμα των σχέσεων της Ρωσίας με πολλές από τις χώρες που θεωρεί ότι ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της και που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για να τις επαναφέρει στη σφαίρα επιρροής της. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να συνεχίσουμε τις πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο διατρανώνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα προς τη Ρωσία. Πριν δώσω το λόγο στον Κρίστοφ Λίσεκ, που είναι και ο συγγετής μας για τη Γεωργία, θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπε η Άννα ε, για το προσωπικό της αποστολής και τη στρατιωτική πείρα που έχουν μερικοί από αυτούς. Διαπιστώνουμε λοιπόν στην αποστολή αυτή ότι η διαφορά μεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού σκέλους είναι τεχνητή, πολύ τεχνητή. Και στα θέματα σχεδιασμού αλλά και σε θέματα προσωπικού επιτόπου η σχέση πολιτικού και στρατικού σκέλους είναι πολύ σημαντική. Αυτό το θέμα της συνοριοποίησης είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα αυτό και χρήζει ικανότητες παρατηρητικότητας που είναι περισσότερο αντανακλαστικά των στρατιωτικών. Και οι άρρηκτα συνδεδεμένες ε, πτυχές και η στρατιωτική και η πολιτική είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της αποστολής, γιατί πολλές φορές τις εργασίες μας ε, διαχωρίζουμε με στεγανό τρόπο, αλλά πολύ τεχνικά, το πολιτικό από το στρατικό σκέλος, το πολιτικό από το στρατικό κόσμο. Σίγουρα είναι πολιτική αποστολή, είναι πολιτικό το αρχηγείο, αλλά το γεγονό ότι υπάρχει στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη βοηθάει πολύ την αποστολή και είναι πολύ χρήσιμη και στο, Ρεχόν, στο Τορεχόν κοντά στη Μαδρίτη πήγαμε στο δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγο καιρό και είδαμε ποια είναι η συμβολή τέτοιων αποστολών και σίγουρα η αποστολή αυτή φάνηκε και η συμβολή αυτή φάνηκε ιδιαίτερα στην αποστολή επιτήρησης ε, στη Γεωργία γιατί ακριβώς το κέντρο της τορεχόν έδωσε κάποιες ε, δορυφορικές φωτογραφίες ε, που ήταν πολύ χρήσιμες και πολύ ενδιαφέρουσες. Μερικοί συνάδελφοι διαρωτώνται ακόμη τι γίνεται με αυτή την στρατηγική αυτονομία που διεκδικούμε. Έχουμε δυνατότητα και ικανότητες εμείς οι Ευρωπαίοι, ικανότητες των κρατών μελών γιατί έχουμε συνένεση για την ε, συνεκμετάλλευση των πόρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δορυφορικές ικανότητες και όλες αυτές οι ικανότητες και η κοινή διαχείρισή τους εξυπηρετεί τέτοιες αποστολές. Και σηματοδοτούν την πραγματική προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Ο Ξύστοφ Λίσεκ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η αποστολή της υποεπιτροπής μας στην Γεωργία. Ήταν και προσωπικά για μένα πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, γιατί ήταν και η, επέτειος, η 20η επέτειος ε, των επισκέψεών μου στην ε, Γεωργία. Και μάλιστα μου είχαν πει ότι αν η Γεωργία ήταν στην Ευρωπαϊκή, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσα να κατέβω και στις ε, γεωργικές ευρωεκλογές. Γεωργιανές μάλλον ευρωεκλογές. Ήταν το αστείο που μας έκαναν οι Γεωργιανοί. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω σε αυτά που είπε ο πρόεδρος ε, Ντανζό ότι έχουμε ε, μια πολύ καλή εικόνα ως Ευρωπαίοι στη Γεωργία και πολύ αναγνωρισμένη. Και σίγουρα η πολιτική σύγκρουση και η πολιτική πόλωση είναι πολύ έντονες στη Γεωργία. Αλλά ένα κοινό σημείο μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι η στάση του απέναντι στην αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η θετική του στάση απέναντι στην αποστολή επιτήρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θα ήθελα φυσικά να χαρώ τον ε, νέο επικεφαλής αποστολής για την ανάληψη των καθηκόντων του και να τονίσω, συνάδελφε, ότι ε, ο νέος επικεφαλής θα έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα εξαιτία της ε, στάσης της Ρωσίας και των αποσχιστικών τάσεων της Νοτιού Οσετίας και της Απχασίας, αλλά ε, η κατοχή του ρωσικού στρατού δυσκολεύει ε, την κατάσταση και εμποδίζει την πλήρη διεξαγωγή της αποστολής. Πάντως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να αφιστεί προσπαθειών ώστε να διευκολύνει αυτή την αποστολή και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συνεχίσουμε τα διαβήματα και να υπενθυμίσω και τη συμφωνία του 2008 που θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθεί. Δυστυχώς ε, είχαμε μερικές φορές τα εμπόδια από τον ε, ρωσικό στρατό και μερικές φορές ε, πώς πέρασαν οι πιέσεις και στην οικονομία. Είχαμε μια τέτοια επίσκεψη όπου είχαμε τέτοια μια περίπτωση που μια η Γεωργιανή είχε το σπίτι της χτισμένο στο τμήμα που έλεγχε η Ρωσία και την τουαλέτα της στην ε, περιοχή που έλεγχαν οι Νότιοι Ήταν θραματική κατάσταση. Στο ίδιο το νοικοκυριό υπήρχε τέτοιος ε, διαχωρισμός. Και υπήρχε και ο φράχτης που κανονικά έπρεπε να χωρίσει και ένα νεκροταφείο. Ένα, στη μέση ένα νεκροταφείο ε, και να χώριζε το νεκροταφείο από το χωριό. Ουσιαστικά δηλαδή ε, οι οικογένειες ε, των ε, θυμάτων των όσων ήταν ανταφιασμένοι στο νεκροταφείο δεν είχαν δικαίωμα εξαιτία του φράγματος αυτού να επισκεφτούν τους τάφους των δικών τους. Και παραπανέθηκαν οι οικογένειες γιατί και σε περιπτώσεις που οι οικογένειες ήταν μακριά από τα παιδιά τους ε, δεν είχαν δικαίωμα επισκέψεων συχνά γιατί τα σύνορα άνοιγαν για λίγες ώρες ε, μόνο και μετά έκλαιναν. Είναι πραγματικά μια κατάσταση που έχει και ε, μια ανθρώπινη πτυχή και μια τραγική ανθρώπινη πτυχή. Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την αποστολή γιατί είναι η μόνη διεθνής αποστολή στην περιοχή που λειτουργεί και ο νέος επικεφαλής μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα κάνουμε από πλευράς μας ό,τι είναι δυνατό για να τη στηρίξουμε. Και ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και η Γεωργική Βουλή και την επόμενη ε, και η δική μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποστολή του ΕΛΚ στο, στη Γεωργία θα είναι η 21η μου επίσκεψη στη Γεωργία και φυσικά συμμετέχουμε στην αποστολή παρατήρησης ε, για τις προεδρικές εκλογές. Και ελπίζω οι εκλογές αυτές να γίνουν με βάση τους δημοκρατικούς κανόνες και σε σχετικά ήρεμο κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κριστόφ. Άλλες ε, παρεμβάσεις σχετικά με αυτήν την επίσκεψη στην ε, Γεωργία. Από ό,τι φαίνεται όχι και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση της κυρίας Μαριάννα Κοπά, εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ετήσια έκθεσή μας που αυτή την ε, χρονιά ε, ε, παίρνει ιδιαίτερο βάρος λόγω του, γεγονός, του γεγονότος ότι το Συμβούλιο θα ασχοληθεί το Δεκέμβριο με διάσκεψη κορυφής για τα, με τα θέματα ασφάλειας. Θέλαμε λοιπόν αυτή η έκθεση να αποτελέσει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, επί του θέματος ε, αυτού, αποσαφηνίζοντας βεβαίως δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι κανείς δεν μας το ζήτησε αυτό ε, και εμείς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Είναι προφανές ότι κανείς δεν ήθελε να διαβουλευτεί με το Κοινοβούλιο. Ξέρετε πόσο ε, τα κράτη-μέλη είναι ε, προσεκτικά ή τέλος πάντων κρατάνε με ζηλοτυπία για τους εαυτούς τους αυτήν την δυνατότητα ε, που τους δίνει το πολιτικό του σύστημα. Εμείς αποφασίσαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ε, γιατί βεβαίως διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Βρισκόμαστε ήδη μέσα Σεπτεμβρίου, ούτε τρεις μήνες δηλαδή από το Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουμε δει καμία συγκεκριμένη και ουσιαστική πρόταση και καμία ουσιαστική τροφοδότηση της ε, ε, συζήτησης. Πολλές ιδέες ακούγονται, πολλά κυκλοφορούν ε, βεβαίως ε, υπάρχουν και διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών, αυτό δεν είναι αμεληταίο, αλλά παρόλα αυτά ε, φοβόμαστε ότι η προθέσεις ε, και οι φιλοδοξίες είναι περιορισμένες. Ε, αλλά βεβαίως μπορεί να ρωτηθεί κανείς ε, μέχρι τώρα είχαμε πολλές ιδέες και πολλές εκπεφρασμένες φιλοδοξίες αλλά με μικρά αποτελέσματα. Θα προτιμούσαμε λιγότερα λόγια και λιγότερες φιλοδοξίες και περισσότερα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, εάν καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας μέσα στα χρονικά περιθώρια που μας επιβάλλουν επιβάλλονται ε, μπορούμε να προχωρήσουμε με ε, τον ε, την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Είναι σημαντικό ζήτημα, επομένως γιατί να μην το καταφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει εμείς το Νοέμβριο ε, θα ολοκληρώσουμε ε, την ε, έκθεση αυτή το Νοέμβριο είτε παρουσία της είπα της εκπροσώπου είτε χωρίς αυτήν δεν έχει σημασία. Εμείς θα υποβάλουμε λοιπόν τις προτάσεις μας και επομένως θα έχουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο στο Συμβούλιο θα έχουν άλλο ένα έγγραφο. Μαριλένα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε είναι σημαντικό να έχουμε ολοκληρώσει την διατύπωση της θέσης μας μέχρι τον Νοέμβριο και θα είναι κρίμα να μην μπορέσει να έρθει η κυρία Άστον, η Λέδη Άστον. Έχουμε περάσει από τα διάφορα στάδια σε, στις συζητήσεις για την άμυνα. Θα είναι σημαντικό λοιπόν εκείνη τη χρονική στιγμή να δοθεί ένα ε, καθαρό μήνυμα. σημαντική ευκαιρία για τους ηγέτες της Ευρώπης και για όλους μας να συζητήσουν τον Δεκέμβρη τις ε, προκλήσεις άμυνας που αντιμετωπίζει η Ένωση και τους ε, σπανιότερους πόρους. Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ένωσης ως πάροχο ασφάλειας και ως παγκόσμιο παράγοντα. Για τον λόγο αυτό απεφάσισα να συντάξω ας πούμε κάπως διαφορετική έκθεση με διαφορετική προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά το μορφότυπο της έκθεσης. Έκθεση στοχευμένη στην ε, επικείμενη διάσκεψη κορυφής και γραμμένη σε απλή γλώσσα, ώστε όποιο πολίτη ενδιαφέρεται να μπορεί να τη διαβάσει και να την καταλάβει. λίγους μήνε πριν από τις ευρωεκλογέ βρίσκω ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι έχει σημασία η άμυνα και μάλιστα ακόμα περισσότερο τώρα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει οικονομική κρίση και αυξημένη αστάθεια στην, ε, στις γειτονικές της περιοχές. Έχω λοιπόν συντάξει την έκθεσή μου γύρω από τα τρία βασικά θέματα που περιλαμβάνει και η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους παραγοντές προσπάθησα να κατανοήσω ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να προσεγγίσουν οι αρχή και κυβερνήσεων. Έκανα μια προσπάθεια να μην προχωρήσω πέραν αυτών και δεν ε, ασχολήθηκα με όλες τις πτυχές της ε, κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι επί του παρόντος δεν θα είχε νόημα να υπησέλθουμε σε όλες τις ε, πτυχές της πολιτικής αυτής και θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει να καθορίσουμε το ρόλο που θα παίξει το Κοινοβούλιο μέσα στη διαδικασία αυτή. Έστω και αν δεν το ζητάνε το ρόλο αυτό όπως είπε και ο Πρόεδρος μας. Για το λόγο αυτό σας παρακαλώ να περιορίσετε επίσης τις τροπολογίες σας αυτά τα πράγματα που έχουν πραγματική σημασία για την επικείμενη συζήτηση, ώστε να μην χάσουμε τη στόχευση για το τι διακυβεύεται. Βεβαίως μπορεί να πει κανεί πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όμως όλα. Νομίζω ότι αν είναι απλούστερη η μορφή θα είναι και πιο ε, ισχυρό το μήνυμα. Αναγνωρίζω και το πράττω και στο κείμενό μου ότι δεν είναι εγχείρημα ενός προσώπου, αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία εντάσσεται μέσα και σε άλλες εκθέσεις, όπως ε, της Άννας και της Μαριέτας Γιαννάκου. Και πρόσφατα σχετικά Σπάσκο, Ντάβιτ και Κέλλερ. Αυτές οι εκθέσεις όλες αποδίδουν τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιμέρους θέματα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και βεβαίως δεν έχω καμία επιθυμία να τις αγνοήσω. Αντιθέτως, Πιστεύω ότι η έκθεσή μου αποτελεί μια σύνθεση αυτών των θέσεων. Δεν επιθυμώ να παρουσιάσω την πολιτική θέση ενός πολιτικού σχηματισμού, αλλά να ξεπηδήσει από το Κοινοβούλιο ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Στοχεύω λοιπόν στα πιο σημαντικά μηνύματα. Την ίδια προσέγγιση θα ακολουθήσω και με την έκθεση του Μιχαήλ Γκάλερ για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση για την άμυνα που είναι το άλλο θέμα που θα συζητηθεί στη διάσκεψη κορυφής. Εγώ κράτησα το τμήμα αυτό του σχεδίου εκθέσεώς μου περιορισμένο, με λίγες μόνο γενικές δηλώσεις και η δική μου πρόταση προς τον Μιχαήλ Γκάλερ είναι να συντονιστούμε και να συντάξουμε ίσως κάποιες τροπολογίες μαζί, αν δέχεται, όταν θα ε, ολοκληρώσουμε και την εργασία μας, Τώρα να έρθω στην δική μου έκθεση. Δεν θέλω να σας κουράσω, έχετε το κείμενό μου, δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες. Ορισμένα κύρια σημεία, τι αναμένουμε πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ασφαλώς δεν αναμένουμε οι ηγέτες να συζητήσουν τεχνικές ρυθμίσεις, αλλά να δώσουν καθαρές πολιτικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της ΚΕΠΑ και για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ωστόσο, δεν θέλουμε άλλη μια καινή περιεχομένου συζήτηση με υποσχέσεις που δεν πρόκειται να τηρηθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρειάζεται πρωτίστως και γι' αυτό νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε υψηλές τις φιλοδοξίες μας, να ξεκαθαρίσει το στρατηγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι προσπάθειες αυτές θα υλοποιηθούν και να ζητήσει από την ύπατη εκπρόσωπο τέλη του 2014 να υποβάλει νέα στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη το νέο στρατηγικό περιβάλλον, να καθορίσει προτεραιότητες και ιδίω για την άμεση γειτονιά μα. ώστε να αυξηθεί η ορατότητα και αποτελεσματικότητα της ΚΕΠΑ, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να ενταχθεί καλύτερα στο στρατηγικό πλαίσιο. Από τη μεριά του οι χώρες μέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν πληρώς τα όσα ήδη περιλαμβάνονται στις συνθήκε τη Ένωση και βεβαίω και την διαρκή διαθρωμένη συνεργασία. Έχει έρθει η ώρα να δεχθούμε ότι δεν θα είναι έτοιμες και οι 28 χώρες μέλη να προχωρήσουν αποφασιστικά μπροστά στην ασφάλεια και άμυνα. Όμως κανεί κανείς δεν επιτρέπεται να εμποδίσει τους άλλους που επιθυμούν. Αυτό που για μένα μετρά περισσότερο είναι όλες οι πρωτοβουλίες να έχουν μια ορατή, αναγνωρίσιμη ευρωπαϊκή διάσταση και να μην υπονομεύουν με κανένα τρόπο την Ένωση και το ρόλο της ανά τον κόσμο. Η δική μου σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι να δώσει ξεκάθαρε συστάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης για την ε, ΚΕΠΑ. Ένα κέριο θέμα είναι η χρηματοδότηση των αποστολών της ΚΕΠΑ, των μάχημων μονάδων και η ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους χώρες μέλη έχουν, το γνωρίζουμε, σημαντική επίπτωση στην επιθυμία τους να συμμετάσχουν. Γι' αυτό χρειάζεται αναθεώρηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών και να δοθεί να μελετηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, εγώ κάνω ορισμένες συστάσεις στην παραγραφό μου 38, ζητώντας ιδίως την πολιτική ενίσχυση για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες του ΕΟΑ και με ένα ορίζοντα του 2025 μαζί και με ε, ένα ειδικό τίτλο για την ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία. Όλα αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν τον Δεκέμβρη, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία που να οδηγήσει σε μια κοινή ανάπτυξη της ε, ΚΕΠΑ στην Ευρώπη. Γι' αυτό ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσει από τώρα ποια συνέχεια θα δοθεί στον προβληματισμό του να φτιάξει ένα οδικό χάρτη με ορόσημα, με τακτικές εκθέσεις και να περιλάβει τα θέματα ε, της άμυνας και της ασφάλειας τακτικά στις ημερήσεις διατάξεις του. Αρκούμε σε αυτά και αναμένω ε, τα σχόλιά σας. Euh. Σας ευχαριστούμε Μαρία Λένα. Είμαι ο σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή, για την γνωμάτωση αυτή. Αλλά δεν έχω σχόλια. Ούτε έχω τίποτα να προσθέσω. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό καταρχάς να έχουμε μια έκθεση που θα είναι περιεκτική, συνοπτική, με ισχυρά πολιτικά μηνύματα γιατί δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε θέματα που έχουμε αναλύσει πολύ λεπτομεριακά τα προηγούμενα χρόνια. Καλό είναι να εστιαστούμε στα πιο στεναρά μηνύματα που θα πρέπει να στείλουμε προς το Συμβούλιο, στα πιο ηχηρά μηνύματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ουσιαστική υλοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της Λισαβόνας, αυτό είναι ένα θέμα που μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θα πρέπει να υπερισχύσει. Φυσικά γνωρίζουμε τις πολιτικές και τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται και με τις ε, δομές, ε, δομή σχεδιασμού και διεξαγωγής των αποστολών και επιχειρήσεων ε, που θέλουμε να βελτιωθεί, το θέμα των battle groups, των μάχημων δυνάμεων ή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικό να αναφέρονται ρητά στην έκθεσή μας και να επιμείνουμε στις διεκδικήσεις μας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στη συνέχεια τα κράτη είναι κυρίαρχα και θα κάνουν μεταξύ τους ε, διάφορες συνεννοήσεις, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι συζητήσεις θα κολλήσουν ως συνήθως σε ορισμένα από αυτά τα σημεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να υποτιμήσουμε ή να ε, μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας για το θέμα αυτό ή τις αξιώσεις μας. Αυτά δεν έχω άλλα σχόλια γιατί η ομάδα μου πραγματικά στερνίζεται και τις προτάσεις και τις διαπιστώσεις που αναφέρει η στην έκθεση και μπορεί για κάποια θέματα λεπτομέρειας να υποβάλουμε κάποια σχόλια αλλά σίγουρα οι βασικοί προσανατολισμοί μας βρίσκουν σύμφωνος και σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική σας έκθεση. Ο κύριος Ντάφ τώρα, από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κοπά για το καταπληκτικό σχέδιο έκθεσης που είναι συγκροτημένο, ε, ορθολογικό, μεστό και μετριοπαθές ως προς τις φιλοδοξίες του. Ως προς την ε, διεύρυνση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά στους ε, καιρούς που ζούμε η μετριοπάθεια είναι πολύ συνετή. Σωστά εστιάζεστε στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, που θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και στρατηγικής ή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερος που το Συμβούλιο βρήκε επιτέλους σε λίγο χρόνο στο πρόγραμμά του να αφιερωθεί στα θέματα αυτά. Επιτέλους ε, βρήκε χρόνο και για κάτι άλλο πέραν της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Φοβάμαι ότι η, ότι στόχη στόχοι του πρόεδρου Βαρνομπόη είναι ακόμη αόριστη, ασαφής και μάλλον περιορισμένη. Και εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προκειμένου να διευκρινιστούν και να ενισχυθούν ε, οι στόχοι αυτοί και να πούμε τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής. Θα έδινε ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Γνωρίζω ότι και εσείς το έχετε περιλάβει στο, στο πρόγραμμα, αλλά για παράδειγμα το θέμα της συμμετοχής του Γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Ράσμουσεν, στην ε, διάσκεψη κορυφής θα συνέβαλε στο να εστιαστεί καλύτερα προσοχή των Πρωθυπουργών και Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων σε αυτό το θέμα. Γιατί ο κύριος Ράσμουσεν ε, ε, πολύ εύγολοτα ε, θα μιλήσει για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στρατιωτικά, ακόμη και στους καιρούς των περιορισμένων ε, αμυντικών δαπανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαριλημμένο ζήτησε λευκή βίβλο για την ασφάλεια και άμυνα. Θα πρέπει τώρα να αντιληφθούμε ότι δεν θα γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Αλλά αν μη τι άλλο θα πρέπει να προωθήσουμε κάποια κοινή προσπάθεια και γιατί όχι και ένα κοινό γνώμονα για τις ε, εθνικές ε, αναθεωρήσεις ε, της ασφάλειας και άμυνας της κοινή πολιτικής που θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Και αν δεν διαρωτηθούν πώς θα ενισχύσουν τις ε, όλο και ξεσθενημένες στρατικές ικανότητες που έχουμε, τουλάχιστον θα πρέπει να δώσουν μια συγκροτημένη απάντηση σε θέματα που είναι πολύ σοβαρά και που όλοι αντιμετωπίζουμε. Επίσης, συμφωνούμε με την εισηγήτρια που θέλει να πατήσει τον γκάζι και να φέρει τα πιο πρόθυμα και στρατικά ικανά κράτη-μέλη να επιταχύνουν και να ενισχύσουν την δική τους ολοκλήρωση ως προπομπό μιας προσπάθειας που θα καταλήξει σε μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λέζινγκ που είναι ε, εξ της ε, ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κυρία Κόπα. Είπατε ήδη στην αρχή της παρεμβάσεώς σας ότι δεν ε, σκέπτεστε να εφεύρετε ξανά από την αρχή τον τροχό, αλλά ότι εντάσσετε την έκθεσή σας μέσα σε μια πορεία και άλλων εκθέσεων. Η έκθεση άλλωστε προβαίνει σε συστηματική καταχώρηση απαιτήσεων για την ενίσχυση της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που ήδη έχουν δηλωθεί και είναι γνωστό ότι για την δική μας πολιτική ομάδα εμείς έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες ε, της εκθέσεως ανακοινώνω ότι θα υποβάλουμε δική μας εναλλακτική έκθεση μειοψηφία. Μένουν ωστόσο ορισμένες ερωτήσεις. Πρόσεξα, κυρία Κοπά, ότι και αυτή η συστηματική σας κατάταξη, σε κλάστερ δηλαδή, ακολουθεί την συστηματική κατάταξη του εγγράφου προτάσεων του γαλλογερμανικού για το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν όλα αυτά συναρμόζονται πολύ ωραία από ό,τι βλέπω. Ερωτήσεις. Στο άρθρο 10 εσείς προχωρείτε σε μια επικαιροποίηση της, ε, ζητείτε μάλλον μια επικαιροποίηση της στρατηγικής συστηματικά δεν είναι τόσο σαφές για μένα πώς είναι δηλαδή δυνατόν να ε, περιγράφετε πρώτα το συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να προκύψει από αυτή τη νέα διατύπωση και μετά να προχωρείτε σε μια περιγραφή της προσπάθειας υλοποίησης της στρατηγικής. Η λογική δική μου θα έλεγε ότι πρέπει να πάει ανάποδα. Ίσως όμως μπορείτε αν θέλετε εσείς να μου το εξηγήσετε πώς δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνετε το δεύτερο βήμα πριν να κάνετε το πρώτο. Και μια καθαρή διευκρινιστική ερώτηση. Στο 19, στο άρθρο 19 ζητείτε, αναφέρετε μάλλον, την ανάγκη να υπάρχουν μόνιμες μάχημες δυνάμεις. Τι ακριβώς εννοείται. Άρα θα σταματήσει αυτό, αυτή η μέχρι τώρα ισχύουσα αρχή της διαδοχικής εναλλαγής, αλλά θα έχουμε δηλαδή μια, ένα πραγματικό στρατό μόνιμο. Ε, ε, πώς, πώς θα πρέπει να ερμηνεύσω αυτή την ε, αξίωση που προβάλλετε εσείς ε, στο άρθρο 19 της εκθέσεώς σας. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου όσον αφορά, να πω δύο λόγια όσον αφορά τη διάρθρωση της ε, έκθεσης. Αναφέρθηκε σε αυτό και η κυρία Κοπά. Είναι όντως, ε, υπάρχουν κάποιες αναλογίες με άλλες ε, εκθέσεις γιατί ούτως ή άλλως ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο και ακολουθεί ε, την, ε, τα τρία στοιχεία, τα, τα, τα, τρεις πτυχές που έχει ακολουθήσει και το Συμβούλιο. Είναι το, η πρώτη πτυχή που αφορά την ορατότητα, δεύτερον τις δυνάμεις, τρίτον την τεχνολογία. Ακολουθούν όλοι την ίδια διάρθρωση ούτως ή άλλως ο κύριος Βανόρντεν τον οποίον βλέπω να μην κρατιέται από τον ενθουσιασμό του εν αυτού του Συμβουλίου. Well, ε, βεβαίως ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα υπέρ της εθνικής ε, ε, ε, απόφασης όσον αφορά τη, και της εθνικής κυριαρχίας όσον αφορά ε, τα θέματα της ασφάλειας των στρατών κτλ. Τέλος πάντων γνωρίζετε γιατί είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια η θέση μου όσον αφορά ε, την ΚΕΠΑ. Ε, πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο κινείται και προωθείται από την ε, θέληση, τη βούληση να υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση αλλά δεν θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ξεχωριστές δομές. Εγώ πάντα έλεγα ότι εάν θέλει να γίνει η Ευρώπη ένα αντίπαλο δέος πραγματικό για τις Ηνωμένες θα πρέπει ε, να ενισχύσει τις πολιτικές και όχι τις στρατιωτικές ε, δομές της. Ε, όσον αφορά την ίδια την έκθεση, την διάβασα, τη διάβασα προσεκτικά και βεβαίως μπορεί κανείς ξεκινώντας από μικρά στοιχεία να δει στοιχεία με τα οποία δεν μπορεί να συμφωνήσει ή μπορεί να συμφωνήσει. Εν πάση περιπτώσει την δημιουργία ενός ε, σταθερού στρατηγίου. Η ε, κυβέρνηση της, ε, ένα μόνιμο στρατιωτικό επιχειρησιακό στρατηγείο. Η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας αντιτίθεται σε αυτό. Ε, όσον αφορά την ε, ΚΕΠΑ ε, και όσον αφορά την δημιουργία μονίμων δομών είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, ούτως υπάρχουν ήδη κοινέ επιχειρήσεις μεταξύ των συμμάχων και μάλιστα όχι μόνο μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η μόνιμη δομή ε, ε, επίσης η εναρμόνιση των ε, κύκλων στους, στις 28 χώρες, όχι αυτό, ούτως ή άλλως είναι εθνική δικαιοδοσία και εν πάση περιπτώσει εν σε επικαλύπτει τις ήδη υπάρχουσες δομές του ΝΑΤΟ. Τώρα όσον αφορά τις μάχημες δυνάμεις και τα μόνιμα και, και τις μόνιμες δυνάμεις εκστρατείας ούτε με αυτό συμφωνούμε. Ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθεί επιπλέον στρατιωτική ικανότητα και βεβαίως ελοχεύει και ο κίνδυνος ε, κάποιες χώρες να πληρώσουν διπλά. Ε, γιατί ε, στο τέλος αυτές είναι δυνάμεις οι οποίες ήδη υπάρχουν ε, στις ε, χώρες και μάλιστα κανείς δεν μπορεί να ανακατευτεί με το στρατό του κάθε έθνους και μετά αφού θα έχει πληρώσει λοιπόν για αυτή τη δημιουργία των ομάδων θα πρέπει να ξαναπληρώσει για την κοινή λειτουργία των μονάδων αυτών. Βεβαίως το κυρίαρχο πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε η βούληση ούτε η πολιτική θέληση να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές ε, δυνάμεις με τρόπο ουσιώδη που θα σήμαινε κάτι δηλαδή. Ε, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν επιπλέον ε, προσέγγιση, αυτοί οι οποίοι αγαπούν ήδη την Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία, βλέπουν όλα αυτά, όλες αυτές τις ε, ε, προτάσεις ε, σαν όλες αυτές τις προτάσεις στα πλαίσια της ΚΕΠΑ τα βλέπουν σαν επικάλυψη των ήδη ισχνών μέσων που υπάρχουν και επομένως καταλαβαίνετε ποια θα είναι και η θέση μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η κυρία Κόνμπεργκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια και να χαιρετήσω το σχέδιο έκθεσης που είναι καλά συγκροτημένο, συνοπτικό, μεστό σχέδιο. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. δεν είχαμε αντιληφθεί τη δυνατότητα εφαρμογής της σε μεμονωμένες αποστολές και επιχειρήσεις ε, τη ΚΕΠΑ. Νόμιζα ότι μόνο σε θεσμική συνεργασία μπορούσε να εφαρμοστεί και όχι σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και αποστολές ΚΕΠΑ. Δεύτερον, ε, διαρωτόμαστε ποιος είναι ο ρόλος της ΚΕΠΑ σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει μια στρατηγική ε, σε ό,τι αφορά ικανότητε ικανότητες ε, της ΚΕΠΑ. Θέλουμε μια διευκρίνηση στο σημείο αυτό. Μας άρεσε ιδιαίτερα, μας άρεσε ιδιαίτερα η παράγραφη για τη γειτονία και το θέμα της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των κρίσεων στις γειτονικέ μας περιοχές. Επίσης, ε, θέλουμε περισσότερη πολιτική συνεργασία και χαιρετίζουμε και την πρόταση για το σώμα μη στρατητικών εφέδρων. Να μην ξεχνούμε ότι τι περισσότερε επιχειρήσει και αποστολέ και πάει είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν είναι στρατητικέ. Σε ό,τι αφορά τι μάχημε ομάδε, μάχημε δυνάμει, battle groups, διαφωνούμε ότι είναι πρόβλημα το ότι οι μάχημε αυτέ οι μονάδε δεν χρησιμοποιήθηκαν. Γιατί ο καλό στρατό είναι ο στρατό που δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν θα φτάσουμε μέχρι τα άκρα να το χρησιμοποιήσουμε η χρήση ή μη χρήση των μάχημων δυνάμεων δεν είναι κριτήριο για τη χρησιμότητά τους. Γιατί κάποιος ρώτησε γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν στο Κονγκό για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα στρατηγικά θαλάσσια συμφέροντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΚΕΠΑ όμως πρέπει να σταθεροποιήσει ε, την ασφάλεια και όχι να προωθήσει οικονομικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε ε, γενικώ το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση στο τομέα της άμυνας. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. I think the civilian sector should have priority in this case and, and uh, the... Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στη, στις πολιτικές επιχειρήσεις, στον πολιτικό τομέα ε, προτεραιότητα και καλύτερα να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στον πολιτικό τομέα παρά στον αμυντικό. Alors, pour terminer avec les, les différents groupes et rapporteurs fictifs, Monsieur Terreau. Ensuite, je repasserai la parole à, à d'autres personnes. Mais... Ο κύριος Τέρα, που είναι ο τελευταίος και αντισηγητής, μετά θα δώσουμε το λόγο στους υπόλοιπους ε, ευρωβουλευτές. Συνήθως συμφωνώ με τους συναδέλφους από την ομάδα των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών, αλλά αυτή τη φορά ομολογώ ότι είμαι κάπως πιο αισιόδοξο ε, για την έκθεση. Και θα συνεχίσω στα φιλανδικά. Πιστεύω ότι είναι η γνωμοδότηση αυτή πηγαίνει πραγματικά σε βάθος. Δεν έχω γενικά σχόλια, θα κάνω μόνο ορισμένα ειδικά σχόλια, αλλά σαν μια πρώτη παρατήρηση ήθελα να πω ότι η Φιλανδία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ και για τον λόγο αυτό ίσως έχουμε διαφορετική προσέγγιση στην αμυντική πολιτική από ό,τι έχουν άλλες χώρες. κρίσιμες ομάδες χωρών μπορεί να είναι ε, μπορεί να είναι υπέρ της, ε, ε, της ευρωπαϊκής Πολιτική ασφάλεια και άμυνας, αρκεί να μην ενοχλούν άλλου, βέβαια. Οι στόχοι της έκθεση είναι φιλόδοξοι. Εγώ έχω συμμετάσχει και παλαιότερα σε ειρηνευτικέ αποστολές της Ένωσης. Βρίσκω κρίμα το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι μάχημες ομάδες. Δεν έχουν έτσι λάβει, δεν έχουν παίξει κάποιον κανένα σημαντικό ρόλο. Θα μιλήσω για την ναυτική δύναμη τώρα. Προέρχομαι από χώρα της οποίας περίπου το 90% το εξωτερικό εμπόριο περνά από τη θάλασσα, από θαλάσσιες μεταφορές. Βλέπουμε ότι κόβονται, περικόπτονται οι πόροι των προϋπολογισμών σε όλη την Ένωση. Αυτό το βλέπουμε και στο επίπεδο της Ένωσης και στο εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή όμως μειωθούν οι ικανότητες και η τεχνολογία στον χώρο αυτό, είναι πολύ δύσκολο να επανακάμψει κανείς, να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Στην διάσκεψη κορυφής πιστεύω ότι γνωρίζουν τα πράγματα αυτά και είναι πολύ σημαντικό να λάβουν οι αρχή κατών και κυβερνήσεων πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση για τα πράγματα αυτά για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Πάσκου και Γκάλερ, αλλά θα δώσω πρώτα τον λόγο στην ε, Μαρία Έλενα Κοπά για να σχολιάσει τις θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων και μετά θα ξαναξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Κοπά, για τα σχόλιά σας. Είναι προφανές ε, ότι στην συζήτηση αυτή απεικονίζεται η θέση των πολιτικών ομάδων καθώς και οι φιλοδοξίες τους όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, τον ρόλο της κοινής πολιτικής ασφάλειας ε, κτλ. Κατά αυτήν την έννοια δεν θα ξεκινήσουμε φιλοσοφική ή ιδεολογική συζήτηση αλλά θα προσπαθήσω απλά να απαντήσω στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία θίξατε. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ. Στο Βίλνιους πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση ε, με την, ε, υπό την Προεδρία της ε, Λέδης Άστον όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ακούσαμε λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την ανάγκη συνεργασίας και μας είπαν ότι το ΝΑΤΟ χρειάζεται ε, αυτήν τη συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Βίλνιους λοιπόν τα ξαναλέω πριν από δύο εβδομάδες είχαμε συνάντηση ε, για θέματα ασφάλειας. Ο κύριος είναι λοιπόν ήταν καλεσμένος και μπορείτε να διαβάσετε το λόγο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η συζήτηση που λαμβάνει η χώρα τώρα στο ΝΑΤΟ είναι η εξή. Ζητά το ΝΑΤΟ ισχυρή παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην διεθνή σκηνή, γιατί το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι παντού και δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω και της πολιτικής γειτονίας της ε, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Επομένως, ε, έχουμε έκκληση από το ίδιο το ΝΑΤΟ για πιο στενή συνεργασία. Αυτό ε, καταδεικνύει και το τι συζήτηση γίνεται και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Χιος Βανόρτεν, να σας πω ότι βεβαίως δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ η Λεδιάστον. Α, όχι, ο κύριος Ράσμουσεν ήτανε. Ναι, βεβαίω, ο κύριο Ράσμουσεν ε, ε, ε, εκπροσωπεί τι ιδέε των κυβερνήσεων και τι απόψει των κυβερνήσεων, πολλέ εκ των οποίων είναι οι ειδεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ δεν είπα ότι στην ΚΕΠΑ δεν υπάρχουν κάποιε ιδέε. Δηλαδή, εσεί μα λέτε ότι συζήτησε το θέμα αυτό ο εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ. Όχι, ο κύριο Ράσμουσεν ήταν πρόεδρο. Πρόεδρος. Ναι, είναι ενδιαφέρον, λέει η κυρία Κοπά. Πρόεδρος, νομίζω ότι θα πρέπει να ε, τελειώσει, να ολοκληρώσει η Μαρία Ελένα Κοπά και μετά ε, θα ε, κάνουμε τη συζήτηση. Μετά η συζήτηση. Συνεχίζει λοιπόν η κυρία Κοπά. Ο κύριος Νταφ έβαλε μια ιδέα στο τραπέζι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι με ε, βρίσκει σύμφωνη. Οι ευαισθησίε των κρατών μελών είναι πολλές και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η ε, ε, ανεξαρτησία απόφασης καθενός αυτό που χρειαζόμαστε τώρα, οπωσδήποτε απεγνωσμένα ε, για τη διάσκεψη κορυφής, είναι καθαρά σαφή μηνύματα. Όσον αφορά τώρα αυτή την ομαδοποίηση, τα clusters, ε, Κοιτάξτε, εγώ δεν έκανα κάτι από μόνη μου. Ε, η συζήτηση γίνεται ήδη ε, αναπτυχές. Υπάρχουν τρεις πτυχές στη συζήτηση και θεώρησα ότι για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα έπρεπε να ακολουθήσουμε τον ίδιο ακριβώς μορφότυπο ε, της συζήτησης. Βεβαίως, πέρα από αυτό υπάρχουν, προκύπτουν και ιδεολογικά φιλοσοφικά ζητήματα και αυτό θα περιμένω αυτή την έκθεση έκθεση που προτίθεστε να εκπονήσετε. Ε, η γενικότερη θέση στάση του συμβουλίου είναι ε, χαμηλός βαθμός φιλοδοξιών ας πούμε. Ε, εμείς νομίζω ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει σαν ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη των φιλοδοξιών. όσον αφορά το στρατό αυτό που λέμε είναι ότι ούτως ή άλλως ε, τα κονδύλια υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν ε, για το ζήτημα αυτό. Επομένως ας κάνουμε αυτές τις δυνάμεις ικανές να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Ας προσπαθήσουμε τις δομές που έχουμε να τις χρησιμοποιήσουμε καλά. Ε, στρατηγείο λοιπόν και λευκή βίβλος. Ξέρουμε ποια, είναι, η θέση του Κοινοβουλίου και δεν μπορούσα λοιπόν να αμελήσω ε, αυτά τα δύο στοιχεία. Ξέρω ότι δεν θα περάσουν στη διάσκεψη κορυφής, αλλά δεν είναι δυνατόν εγώ να ε, κάνω ότι δεν είσαμε ποτέ για αυτά και ότι δεν μας απασχόλησαν ποτέ. Κυρία Κρόμπεργκ, Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. η βιομηχανία άμυνας και θα έχουμε άλλωστε και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση Γκάλερ. Είναι ένα ε, θέμα για το οποίο υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδεολογικές ε, απόψεις. Μην λησμονούμε πάντως ότι η, η άμυνα η βιομηχανία άμυνας είναι η μόνη η οποία δεν έχει φύγει από την Ευρώπη και δεν μπορεί να φύγει. Όλες οι άλλες βιομηχανίες μπορούν να πάνε στο Πακιστάν, στην Ινδία, όπου θέλουν. Το θέμα λοιπόν είναι να στηρίξουμε και τη βιομηχανία και αυτούς που δουλεύουν στη βιομηχανία αυτή. Α, θαλάσσια ασφάλεια. Άλλο θέμα. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να ε, αναφερθώ στην προστασία συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, αλλά όταν μιλάμε για πειρατεία, ας πούμε, οπωσδήποτε η θέση μας πρέπει να είναι σαφής. Ε, και νομίζω ότι κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ε, να τα καταφέρουμε. Όσον αφορά την ΚΕΠΑ, πολλοί λένε λένε ότι είναι ένας άλλος τρόπος ε, για ερμηνεία της ε, ε, της συνθήκης λειτουργίας της Λισαβόνας. Όταν μιλάμε για Πέσκο, πολλοί σε, αυτήν, σε αυτό το θέμα αναφέρονται. Εξωτερικά σύνορα. Βεβαίως έχουμε, θέμα, έχουμε παραδείγματα προστασίας εξωτερικών σύνορων. Υπάρχει η Frontex, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά στη χώρα μου, στο Αιγαίο. Η προστασία λοιπόν του θαλασσίου χώρου μπορεί να είναι ε, από αυτούς που ε, εμπορεύονται την ανθρώπινη ζωή και που περνάνε τους μετανάστες ή ε, οτιδήποτε άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχει λοιπόν και πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω. Επιμένω επίσης και σε κάποια άλλα θέματα, τα οποία, ε, σε κάτι το οποίο υπάρχει και στο κείμενό μου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αμέσως. Αλλά βεβαίως είμαστε και υπεύθυνοι για τη γειτονιά μας. Το ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά μας οπωσδήποτε επηρεάζει τους πολίτες μας. Ε, και επομένως θα πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι η άμυνα δεν αφορά μονάχα τα στρατιωτικά ζητήματα, δεν είναι μονάχα στρατοί και στρατιώτες η άμυνα. Είναι, ε, αφορά τους ίδιους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως έστω και αν έχουμε κάποια σημεία διαφωνίας θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξηγήσουμε με τρόπο εξωστρεφή και σαφή τα πράγματα αυτά στο θεματολόγιο των ευρωπαϊκών εκλογών δεν πρέπει να διστάζουμε να μιλάμε και για τέτοια θέματα λόγω της περιουραίουσας ατμόσφαιρας και των ε, χαλεπών οικονομικών καιρών. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ. Ήδη λέχθηκαν πολλά. Θα είμαι σύντομος λοιπόν. να σχολιάσω για τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ Βαν Όρντεν και της ε, εισηγήτριάς μας. Την ερώτηση θα μπορούσαμε να τη θέσουμε και σε ένα παιδί. Είναι λίγο σαν να το ρωτάμε αν προτιμά να αγαπά πιο πολύ τη μητέρα από τον πατέρα. Μεταξύ Πολωνίας, Γερμανίας και Γαλλίας αυτό το εμείς περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, γιατί 22 από 28 χώρες είναι μέλη και του ΝΑΤΟ. Και εμείς δεν μπήκαμε στην συμμαχία με σκοπό να τη διαλύσουμε. Είναι συνειδητή επιλογή των ε, ε, ηγετών μας και οι ηγέτες ε, των χωρών μας δεν είναι άνθρωποι παράνοες παλαβοί και, και όλοι θέλουμε να αποφύγουμε επικάλυψη. Το έχουμε πει και το έχετε ακούσει κι εσείς ε, πολλές φορές. Θέλουμε να αποφύγουμε επικάλυψη των προσπαθειών και κατασπατάληση των ε, εσόδων, σίγουρα. Συμφωνούμε με την ε, κυρία Κοπά ότι η υποεπιτροπή μας πρέπει να δείξει ότι και εμείς είμαστε φιλόδοξοι στα θέματα κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και απαιτούμε από τους ηγέτες μας περισσότερα και όχι λιγότερα. Γι' αυτό και εγώ ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να εμείνουμε στην ανάγκη μιας ε, στρατηγικής αντιμετώπισης της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και θα είναι ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τις περιβόητες αυτές δυνάμει, μάχημες δυνάμεις, υπάρχει συμφωνία ότι μερικές φορές κάποια στοιχεία της κοινή πολιτική ε, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν δίνουν καλή εντύπωση. Γι' αυτό και θα πρέπει στη διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου να ζητήσουμε από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν μια απόφαση ή το ένα ή το άλλο ή να εξασφαλίσουν μηχανισμό λειτουργίας και χρηματοδότησης πραγματικών μάχημων δυνάμεων ή αλλιώς να καθαρίσουμε αυτό το θέμα και να σταματήσουμε τις χαζομάρες. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσκου. θα έλεγα ως προς την έκθεση ότι τελικά ξεπερνάμε ένα πρότυπο συμπεριφοράς που συνήθως είχαμε στο παρελθόν ε, που απλώς περιγράφαμε τι συνέβη πέρυσι δηλαδή, ποιες επιχειρήσεις είχαμε πέρυσι και τελείωσε. Αυτό κάναμε μέχρι τώρα. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μας έκανε να αλλάξουμε αυτό το κανόνα συμπεριφοράς και να το βελτιώσουμε η Μαριαλένα έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια και πραγματικά ε, συμφωνώ, τη στηρίζω πλήρως και ενώνω και εγώ τη φωνή μου σε όσους εγκομίασαν την έκθεση. Τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ πιο γενικά με ορισμένα θέματα. Ξεκινήσαμε με κάποιες προσδοκίες ε, απέναντι στο Συμβούλιο. Μετά είδαμε τι συνέβη και κάπως μετριάσαμε τις ε, προσδοκίες μας ναι, από την ε, Σύνοδο Κορυφής. Θα έλεγα όμως ότι οι προσδοκίες μας θα πρέπει να συνδυαστούν με το γεγονός ε, το, ή με την άποψη του κατά πόσο η Σύνοδος Κορυφής είναι μια διαδικασία. Γιατί αν είναι μια διαδικασία και υποσχεθεί ότι στη συνέχεια θα λύσει τα προβλήματα, θα ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα, τότε θα πρέπει πάλι να αναβαθμίσουμε τις φιλοδοξίες μας και να αφήσουμε αυτά τα πράγματα στο Συμβούλιο έχοντας εμπιστοσύνη ότι αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στη συνέχεια. Ελπίζω να μην είναι η Σύνοδος Κορυφής ε, ένα μεμονωμένο γεγονός χωρίς συνέχεια και το επόμενο ε, παρόμοιο Συμβούλιο να είναι μετά από μία πενταετία. Λοιπόν, πιστούμε ότι θα ξεκινήσει τώρα μία διαδικασία, τότε μπορούμε να έχουμε υψηλές προσδοκίες. Βέβαια, αν δεν δοθεί συνέχεια, αν είναι υψηλέ οι προσδοκίε, εξίσου υψηλή θα είναι και μεγάλη θα είναι και η απογοήτευσή μα. Θα πρέπει το Συμβούλιο να δούμε αν θα ξεκινήσει μια διαδικασία συνέχιση και παρακολούθηση των συζητήσεων που θα ξεκινήσει το Δεκέμβριο. Επίση θα πρέπει και σε επίπεδο επιτροπής και σε επίπεδο επιτροπή ε, ΦΕΤ να συνδυάσουμε όλε αυτέ τι εκθέσει ε, που θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμε για το Συμβούλιο και να κάνουμε ένα το σχέμα όλες αυτές τις εκθέσεις τις σχετικές να κυκλοφορήσει αυτό το ντοσιέ, να το μοιράσουμε σε όσους ε, θεωρούμε ότι έχουν κάποια επιρροή και να το βάλουμε και στο, στην ιστοσελίδα μας και να έχουμε ένα, ένα συγκεκριμένο κατάλογο με τις ε, εκθέσεις μας που είναι σχετικές με το αντικείμενο του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζετε ότι το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να ξεπεράσουμε την κουλτούρα ή την οτροπία ότι ό,τι και να συμβεί οι ΙΠΑ θα μας σώσουν. Ναι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και συνθήκες όπου για τον ΑΒ λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες μας θα πρέπει να έχουμε και ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο αναδίπλωσης, γιατί υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να στραφούν απευθεία στο ΝΑΤΟ. Θα στραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητήσουν από εμά υποστήριξη. Γνωρίζουμε ότι ε, η Φιλανδία προστατεύθηκε από το ΝΑΤΟ καθ' όλη την περίοδο της φιλανδοποίησης. Και έτσι κατέστη δυνατή αυτή η διαδικασία χάρη στην έμεση έστω προστασία του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο θέμα. Ούτως ή άλλως ξεπερνούμε αυτή την οτροπία πια ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σε κάθε περίπτωση θα έρθουν και θα μας σώσουν. Ανεπιφύλακτα και ανεφόρον. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενε εκπλήξεις στον τομέα αυτό. Τώρα, ως προς την πολιτική των δυνάμεων. Έχουμε μια νέα ιεράρχηση και σχετισμό δυνάμεων πια στην παγκόσμια σκηνή. Και ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας της ισχύω. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ε, στους μηχανισμούς της εξουσίας περιλαμβανόταν και ο στρατός. Δεν μπορεί κανείς να πει, ναι, ε, Μονομαχό μαζί σου αλλά με το ένα με το δεξί χέρι πίσω και μόνο με το αριστερό κρατάω το σπαθί και κάνουμε την ξεφασκία. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είναι γεγονός. Ε, θα πρέπει να το αποδεχτούμε και να το συμπεριλάβουμε στις, ε, στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, Τάνια, η σχέση μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής παραγωγής είναι πολύ πιο στενή από ό,τι στο παρελθόν και πολύ εύκολα γίνονται μεταφορές ε, από τον ένα κλάδο στον άλλο. Και αξιοποίηση. Παλιά γινόταν αξιοποίηση του, στρα, του στρατιωτικού σκέλους από το πολιτικό, στο, στο διαδίκτυο για παράδειγμα. Τώρα έχουμε και το αντίθετο. Κάποιοι, κάποια προϊόντα της, της μη στρατιωτικής βιομηχανίας μεταφέρονται στη στρατιωτική. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, να επανεξετάσουμε την ορθωτική γραμμή μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού κλάδου που είναι πιο ρευστή από ό,τι στο παρελθόν. Και τελευταίο σχόλιο και σας υπόσχομαι θα τα ολοκληρώσω. Χθες ήμουν σε μια συζήτηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η αίσθηση που μου δημιουργήθηκε από τη συζήτηση είναι ότι ο κόσμος μας σε σχέση με τον εικονικό κόσμο και ο δικός μας είναι ο πραγματικός κόσμος ουσιαστικά ο δικό μα, ο πραγματικό κόσμο είναι ο εικονικό κόσμο. Γιατί ο πραγματικό κόσμο είναι ο εικονικό κόσμο. Όλα εκεί συμβαίνουν. Πώ λοιπόν θα προσδιορίσουμε την ασφάλεια όταν ένα μεγάλο τμήμα τη ασφάλεια συμβαίνει σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Και είδα εμβρόντιτος ότι Μία Αμερικανίδα χθε στη συζήτηση είπε ότι τα αμερικανικά δικαστήρια δεν έχουν τη γνώση, δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα, τέτοιες υποθέσεις. Ο εικονικός χώρος δεν έχει όρια, είναι σαν το σύμπαν. Είναι προσιτό σε όλους και δεν έχει και κανόνες. Όποιος αδράξει ό,τι περισσότερο μπορεί, το κάνει ανενόχλητα. Όλα αυτά αλλάζουν λοιπόν το πλαίσιο αναφοράς μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μείνουμε στο μέτρο του δυνατού όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα που ναι μεν αποκαλούμε εικονική αλλά παρόλα αυτά είναι πραγματικότητα και ο δικός μας ο πραγματικός κόσμος γίνεται όλο και πιο εικονικός. Ευχαριστώ. Αλλά αυτή ήταν μια εξαιρετικά μια παθιασμένη παρουσίαση του πραγματικού κόσμου. Μικαήλ Γκάλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστεί να επαναλάβω τα περισσότερα από όλα αυτά τα πράγματα. Ως συντονιστής του Λαϊκού Κόμματος θέλω να σημειώσω ότι καταρχήν υποστηρίζω την έκθεση της ε, κυρία Κοπά, τη γενική κατεύθυνσή της δηλαδή, ότι είναι σαφές για μας ότι μπορεί να υπάρξουν κοινά σημεία μιας κοινή πορείας. Έχω ωστόσο να πω το εξής ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε παραπάνω από 8% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και εάν θέλουμε να ασκήσουμε μια κοινή πολιτική που να καταστήσει δυνατό να διατηρήσουμε την ευημερία μας, το προβιωτικό μας επίπεδο, αν θέλουμε να τα διαφυλάξουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε. Όποιος θέλει να είναι soft power πρέπει να μπορεί ταυτόχρονα να είναι και hard power δεν σημαίνει ότι θέλει, αλλά οι κρίσεις έρχονται αυτές πάνω μας. Και οι Αμερικανοί φίλοι μας, ο καινούριος εδώ ανώτατος διοικητής στην Μόνς, είπε πρόσφατα στις Βρυξέλλες ότι βεβαίως πάντοτε δεσμευόμαστε από το άρθρο 5, αλλά οτιδήποτε άλλο σε χαμηλότερο επίπεδο από το άρθρο 5, αν είναι η επίθεση από επίπεδο χαμηλότερο από το άρθρο 5, τότε να φροντίσετε εσείς. Αυτό είπε καθαρά. Δεν θέλω να βρεθώ σε μια κατάσταση που ανακολουθώ μόνο τη γραμμή του ΝΑΤΟ εν τέλει, αν δω την αναγκαιότητα, ας πούμε σε ένα μέρος των Βαλκανίων να, να μπορέσω να εμφανιστώ, ξαφνικά να μου βάλει η Τουρκία ένα βέτο, επειδή είμαι εκτός ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν θέλω ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαρτώμαι από τα τα όχι μια τρίτη χώρας. Δεν μπορώ τότε να απαντήσω στο τουρκικό βέτο στην περίπτωση αυτή, γιατί οι αποφάσει στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται ομόφωνα. Δεν θέλω λοιπόν να έχω να αντιμετωπίσω ένα βέτο τρίτης χώρα. Αυτό είναι μία από τις πτυχέ. Επειδή λοιπόν όλοι δεν έχουμε αρκετά λεφτά, γι' αυτό οι προτάσει σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των προγραμμάτων προμηθειών κλπ. Όλα αυτά είναι προς το συμφέρον όλων και για την εξοικονόμηση πόρων αλλά και για την αύξηση της διαλειτουργικότητας. Ποιος μπορεί να είναι αντίθετο σε αυτά. Αυτά λοιπόν τα βάζω και ως πρόσθετα επιχειρήματα που ενισχύουν την αρχοκοκαλιά της έκθεσης. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κοπά για το σχέδιο εκθέσεω που κατέθεσε. Πολύ ωραία. Να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση. Αυτή ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Αλλά χαίρομαι για το ενδιαφέρον που προκαλεί αυτό το θέμα, αναμενόμενο βέβαια. Τρεις ακόμη συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και μετά θα εξετάσουμε την έκθεση Γκάλερ. Τρεις ομιλητέ και μετά για τη δευτερολογία και τα συμπεράσματα κυρία Κοπά. Η κυρία Κρόμπερκ, μετά η κυρία Λέζιν και μετά ο κύριος Κάμπελ. άγεται και Τζέφρι Όρντεν. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ και τι είπε στο Βίλνιους ο ενώ ο γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ότι το ΝΑΤΟ θέλει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε όμως ε, ταυτόχρονα ότι το βασικό σημείο είναι η Κύπρος, οπότε η θεσμική συνεργασία δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα για το εγγύς μέλλον. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τις δικές της ανάγκες και με βάση αυτές να κρίνει. Σε ό,τι αφορά τις μάχημες δυνάμει, τα battle groups, ναι, κατανοώ το επιχείρημά σας ότι αν δεν τις χρησιμοποιούμε ίσως θα πρέπει να τις καταργήσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε, να χρησιμοποιούνται σωστά. Το θέμα είναι τι θα πει καλή χρήση, σωστή χρήση των μάχημων δυνάμεων. Θα πρέπει να ορίσουμε την καλή χρήση. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τόσα μεμονωμένα κρατικά συμφέροντα και μερικές φορές γίνεται παρερμηνία. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, μάχημες δυνάμεις θα πρέπει να προσδιορίσουμε, να ορίσουμε τον όρο καλή χρήση. Τώρα σε ό,τι αφορά την στρατιωτική βιομηχανία, την αμυντική βιομηχανία, το θέμα δεν είναι μόνο με, μετεγκατάσταση, γιατί και η αμυντική βιομηχανία μπορεί κάλλιστα όπως οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία να μετεγκατασταθεί. Και από ό,τι ξέρω οι Γάλλοι έχουν αναφυγία στην Ρωσία υπάρχει μια διεθνοποίηση και δεν πιστεύω ότι με το επιχείρημα μόνο της μετεκατάστασης για να το αποτρέψουμε θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική στρατιωτική βιομηχανία. Ναι, μεν είναι σημαντική βέβαια για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αυτό το επιχείρημα ίσως θα πρέπει να δούμε πώς θα την προστατεύσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καινοτομία, ένα θέμα που θα εξετάσουμε αργότερα, και αυτό το θέμα είναι προβληματικό αν κλείσουμε ε, την Ευρώπη στις βιομηχανίες και στη στρατιωτική. Σε ό,τι αφορά το Frontex, τη Frontex, νομίζω ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής. Ήταν ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω και το ελληνικό πρόβλημα. Αλλά υπό το πρίσμα της δικής μου πατρίδας Φιλανδίας υπάρχει αντίδραση απέναντι στη Frontex. Δεν θέλουμε να ενισχυθούν οι εξουσίες της ε, γιατί κάθε χώρα που έχει σύνορο θα πρέπει να είναι αρμόδια και υπεύθυνη για τις πολιτικές της. Υπάρχει αυτό το θέμα των εφιών σύνορων, μια πρόταση που ίσως καλό θα ήταν να την αναπτύξουμε περαιτέρω. Αυτά, ευχαριστώ. Merci, <coughs> <coughs> Πρώτα, επανέρχομαι στις έννοιες ιδεολογία και ιδεολογικός κλπ. Δεν συζητούμε ιδεολογίες εδώ, αυτά τα κάνουμε ίσως σε σεμινάρια φιλοσοφίας. Μάλιστα έρχονται και θαυμάσιοι φιλόσοφοι από τη χώρα μου και συνιστώ να τους διαβάσετε. Αυτό που συζητούμε εδώ έχει και συγκεκριμένες επιπτώσεις, πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις και μάλιστα στους προϋπολογισμούς. Για αυτά τα πράγματα συζητούμε μεταξύ άλλων. Γι' αυτό έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Εάν ο κύριος Ράσμουσεν έρχεται και ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο το ΝΑΤΟ, αυτό το κάνει βεβαίως και για δημοσιονομικούς λόγους, για λόγους προϋπολογισμού. Υπό την ηγεσία των Ενωμένων Πολιτειών δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει χρηματοδοτικά όλες αυτές τις αποστολές απέναντι στον Αμερικανικό λαό και γι' αυτό ζητεί τη συμβολή των Ευρωπαίων. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Κύριε Πάσκου, ωραία και καλά αυτά που είπατε. Αυτά που αναφέρατε τώρα για τον Ευρωπαϊκό στρατό ως συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ σε εμά τους αριστερούς δεν μας αρέσουν, αλλά κάποιοι άλλοι αριστεροί τα συζητούν. Θεωρώ ότι πρόκειται για ψευδεστήσεις. Βρισκόμαστε μέσα σε μια στρατηγική συμμαχία και όλες οι στρατηγικές φιλοδοξίες των ΗΠΑ θεωρούνται συμπλήρωμα του ΝΑΤΟ και στην πραγματικότητα πρόκειται ωστόσο μόνο για τη χρηματοδότηση. Το θέμα που έθεσε η κυρία Κρόνμπεργκ, το επαναφέρω και εγώ, σε ό,τι αφορά την εξωτερική μεθόριο, δεν μπορούμε να εξετάζουμε τις εκθέσεις ξεχωριστά, πρέπει να τις συζητούμε συνολικά. Η κυρία Γκόμες την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια είπε ορισμένα πράγματα και μάλιστα πολύ ξεκάθαρα. Είπε ότι η θαλάσσια στρατηγική της Ένωσης οφείλει να εξυπηρετήσει και τον σκοπό της προστασίας των θαλάσσιων συνόρων της Ένωσης ανά τον κόσμο. Ρωτώ εγώ, πού βρίσκονται αυτά τα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης, πώς είναι δυνατόν να φανταστώ ότι οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει τα σύνορά της, τα θαλάσσια μπροστά από τη Σομαλία. Είναι πράγματα αυτά τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν για το μέλλον. Κάτι που μου φαίνεται αξιοσημείωτο και σας συγχαίρω για την εκθεσή σας εν προκειμένου κυρία Κοπά, διότι όταν συζητεί κανείς επιμακρών για μια υπόθεση, τότε αποκομίζει κανείς πολύτιμα συμπεράσματα. Ο κύριος Γκάλερ εξήγησε με λίγα λόγια πολύ καθαρά τη λειτουργία της στρατιωτικής πολιτικής. θέλει να προστατεύσει την ευρωπαϊκή ευημερία με soft power και αν χρειαστεί και με hard power. Αλλά το είπατε πολύ καθαρά αυτό. Και νομίζω ότι σωστό είναι να βγούμε και να τα πούμε αυτά στον κόσμο, στους πολίτες, ε? να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Και έρχομαι και στην ιδέα του κύριου Πάσκου. Τη βρίσκω πολύ καλή. Δηλαδή εκθέσεις αυτές να δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα. Διότι θεωρώ ότι οι στρατηγικές, οι στρατιωτικοπολιτικές στρατηγικές της Ένωσης δεν είναι αρκετά γνωστές στους πολίτες και ούτε συζητούνται αρκετά. Χαίρομαι λοιπόν που επιτέλους διευκρινίζεται και περί τίνος πρόκειται με αυτή την Αταλάντη. Είμαι τέσσερα χρόνια στην υποεπιτροπή αυτή και είχαν πει τότε «Α, θέλουμε να προστατεύσουμε μοναχά τα πλοία τα οποία μεταφέρουν επιστηστική βοήθεια». Κάπου είχε καταληφθεί αυτή η επιχειρηματολογία. Τώρα, τώρα πια μας λένε καθαρά ότι Πρόκειται για προστασία οικονομικών συμφερόντων. Πρόκειται για προστασία της ασφάλειας προμήθειας ενέργειας, την οποία εξασφαλίζουμε στρατιωτικά και ούτω καθεξής. Παρατήρηση του κ. Γκάλερα χωρίς μικρόφωνο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι στρατιωτικές αποστολές αυτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Χαίρομαι λοιπόν που στη συζήτηση αυτή δεν συζητήσαμε ιδεολογικά και θέλω να επανέλθω πάλι σε μια ιδέα του κυρίου Πάσκου, δηλαδή να εξηγήσουμε τα πράγματα αυτά στον κόσμο, στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να συζητηθούν και τουλάχιστον οι άνθρωποι να ξέρουν τι συμβαίνει εδώ, γιατί και πώς. Και μπορούν, εν πάση περιπτώσει, έτσι να αποφασίσουν αν τα θέλουν αυτά τα πράγματα στο μέλλον ή όχι. Ε, ε, τώρα θα πρέπει να ρωτήσουμε και τον κύριο Γκάρλ, θα περιμένουμε κάτι μετά την Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει, Πρόεδρος, να υπενθυμίσω ότι ούτως ή άλλως ε, και οι συζητήσεις που έχουμε και οι εκθέσεις και οι συζητήσεις των εκθέσεων είναι δημόσιες, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους πολίτες να διαβάσουν ή να μας ακούσουν. Ε, και βεβαίως εμείς ως Ευρωπαίοι βουλευτές έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και συζητάμε για τα θέματα αυτά. Και εσείς κυρία Λέζινγκ αν θέλετε μπορείτε στη δικιά σας εκλογική περιφέρεια να οργανώσετε συζητήσεις για την κοινή πολιτική ασφάλεια. Ε, γιατί και η κυρία Κοπά το είπε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι πολίτες μας για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμβαίνει με την άμυνα. Το είδαμε και στην περίπτωση της Λιβύης, του Μαλή, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ενδιαφέροντα ζητήματα για την, για την κοινή γνώμη. Και ο ρόλο μα είναι να ε, συζητάμε για τα θέματα αυτά όσον αφορά την επιχείρηση Αταλάντη. Να σα πω ότι δεν υπήρξε ποτέ κρυφός στόχος της επιχείρησης Αταλάντη προστασία εμπορικών, η προστασία των εμπορικών πλοίων που περνούν από την περιοχή αυτή δεν αφορά μονάχα προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η θαλάσσια προστασία προσφέρεται σε όλα τα ε, πλοία τα οποία περνούν από την ε, περιοχή αυτή. Ε, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως η επιχείρηση Αταλάντη προσπαθεί να μην μπλέξει με πλοία τα οποία έχουν ήδη στρατιωτικούς ε, στα, στα, στο, προσωπικό τους αλλά από την άλλη πλευρά ε, και είναι σαφής ο στόχος αυτός η επιχείρηση Αταλάντη θέλει να προστατεύσει όλα τα πλοία που περνούν από την περιοχή. Ο κύριος Κάμπελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σαφής και καλογραμμένη, αλλά νομίζω ότι μας δημιουργεί μεγάλη κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ κακή ο προσανατολισμός ε, είναι ε, πρώτες κινήσεις προς, ενιαία, ενιαίο στρατό και νομίζω ότι ε, καλό θα ήταν να το πείτε ξεκάθαρα και όχι να το κρύβετε κάτω από άλλες παραγράφους και άλλες ιδέες. Θα πρέπει να το πείτε ξεκάθαρα, να το παραδεχτείτε. Ναι και το ΕΛΚ ε, το ίδιο πρεσβεύει. Βλέπω ότι ζωήρεψε ξαφνικά η υποεπιτροπή και ασχολείται πλέον με θέματα που σχετίζονται με τη συνθήκη λειτουργία της Λισαβόνας αφού έχει περάσει από διάφορα άλλα θέματα. Ε, τώρα ε, γίνεται λόγος ε, για το Συμβούλιο Ασφάλειας, ε, γίνεται λόγος για διαρθρωμένο διάλογο για τα θέματα αυτά. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα λόγο να ανακατευτεί με αυτά τα πράγματα αν τώρα όλο αυτό το θέμα για τις επιπλέον επενδύσεις ή ε, για τα ταμεία τα οποία έχουν αδειάσει στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους οργανισμούς και επομένως θα πρέπει να βάλει το, χέρι στην τσέπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι ε, πράγματα πολύ, ε, τα οποία πρέπει πολύ προσεκτικά να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τώρα αυτά τα battle groups, ε, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ομάδες, θα πρέπει να χυθεί αίμα ε, όλες αυτές έτσι οι πολύ ακραίες ε, διατυπώσεις, λες και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο σε μερικούς μήνες, όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, όλα... ναι, αυτό είναι model thinking. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουν ε, από τα εθνικά κράτη ε, ε, οι πολίτες μας. Θέλουν οπωσδήποτε εθνική κυριαρχία. Παρατηρήσεις εκτός μικροφώνου. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο εξώτημος συνάδελφος εδώ. Νομίζω ότι ο στόχος Νομίζω ότι αυτή η έκθεση ε, απομακρύνει ακόμα περισσότερο την ε, Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν ε, τα πράγματα μέσα σε μία μέρα. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα συμβεί. Θα απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο εάν επιμένετε σε αυτές τις φεντεραλιστικές φιλοδοξίες. συζητήσεις εκτός μικροφώνου. Πρόεδρος. Για να... να ολοκληρώσουμε. Καταρχήν, ε, ε, κατά τη γνώμη μου κάνετε ερμηνεία πολύ παρατραβηγμένη της έκθεσης ΚΟΠΑ και ε, της αποδίδεται προθέσεις που δεν έχει. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις Ε, ε, ε ούτε και στη Γαλλία δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ένα ευρωπαϊκό στρατό που θα ηγείται ένας ε, γραφειοκράτης Ευρωπαίος, ένας ευρωκράτης. Αλλά δεν θα σας πείραζε ένας ε, αμερικανοαγγλικός στρατός ε, που ο ήταν ένας ε, γερουσιαστής. Άλλωστε η ανεξαρτησία που διεκδικείται για την Ευρώπη φαίνεται ότι χάνεται όταν μιλάτε για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι επιχειρήσει των Αμερικανών που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια οδηγούν σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις και συμπεράσματα. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην έκθεση ΚΟΠΑ και να τη διαβάσουμε, αυτά που λέει και να μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να τις αποδίδουμε τέτοιες προθέσεις και διαστάσεις που δεν έχει. Άλλωστε αυτά που λέει η έκθεση περιχαρακώνονται και στη συνθήκη. Μιλάμε για τις διατάξεις της συνθήκης και μπορείτε να είστε κατά της συνθήκης, αλλά έχει κυρωθεί αυτή η συνθήκη. Μετά ο καθένας είναι κυρίαρχος να καθορίσει τη θέση του, αλλά ε, εργαζόμαστε με μία συνθήκη που έχει κυρωθεί και όχι με εφάνταστες ε, θέσεις. Ο κύριος Βανόρδεν, φυσικά είμαι κατά της, ε, θα ήμουν κατά της συνθήκης Λισαβόνας. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα πια και θα πρέπει να την αποδεχτούμε. Μάικλ, μίλησε για τα Βαλκάνια. Μην ξεχνάς ότι οι δύο αποφασιστικές ε, επεμβάσεις στα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια έγιναν από το ΝΑΤΟ. Μην το ξεχνάς. Επανέρχομαι τώρα σε αυτά που αναφέρθηκαν για τον κύριο Ράσμουσαν. Δεν θέλω να κυλιδώσω τη φήμη του σε καμία περίπτωση αλλά είχε έρθει και στην Επιτροπή μας σχετικά πρόσφατα, θυμάμαι καλά. Και ως συνήθως, όταν μιλά σε ακροατήριο ευρωπαϊκό, ε, λέει αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Ε, παραλαμβάνει κάποια μάντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ωραία λόγια και το έκανε και στο Βίλνιους. Είναι ευγενικός άνθρωπος ε, και αυτό περιμένουμε από έναν ε, ευγενικό κύριο. Θέλεις δηλαδή να πιστέψουμε, Τζέφρι, ότι ο Ράσμουσεν δεν εννοεί αυτά που λέει. Και θα πρέπει να, να πιστέψω αυτά που δεν λέει και όχι αυτά που λέει. Τι εννοείς. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Η έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν περισσότερη δράση δεν είναι κάτι καινούριο. Ούτε είναι κάτι που οφείλεται στη μεταστροφή των Αμερικανών προς την Ασία, η μετατόπιση του ενδιαφέροντων των Αμερικανών. Τα τελευταία 60 χρόνια ακούγεται αυτή η έκκληση, η κραυγή προς τους Ευρωπαίους να κάνουν περισσότερα. Μας λέτε επαφιόμαστε στους Αμερικανούς. Όχι, φυσικά και όχι. Και, και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν πυρηνικό όπλο. Σίγουρα δεν θα επαφεθούμε πλήρως στους Αμερικανούς. Δηλαδή, αν λίμωνο. Ε, βλέπω ότι υπάρχει ένας έμεσος εδώ αντιαμερικανισμός. Φαίνεται ότι αυτή είναι η λανθάνωσα τάση ε, στη συζήτηση. Ο Ράσμους, ενώ τα μίλησε με πολύ ευγένεια και αυρότητα στο Βίλνιους, ναι, με ε, απευθυνέ στις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν περισσότερα, αλλά στο τέλος είπε, όσο ταξιδεύουμε θα πρέπει να μην προσπαθούμε να εκτροχιάσουμε τους άλλους από την πορεία τους με παρόμοια σχέδια και επικάλυψη. Δεν έχουμε χρήματα για κάτι τέτοιο, ούτε και φορολογούμενοι έχουν την υπομονή για κάτι τέτοιο. Συνεργασία λοιπόν και όχι επικάλυψη. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε. Και εσείς ως Ευρωβουλευτές θα έχετε αποφασιστικό ρόλο για να ελοποιήσετε κάτι τέτοιο. Αυτά είναι που υποράσμουσε στο Βίλνιους. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα το οποίο μου είναι ιδιαίτερος προσφυλές και χαίρομαι όταν έχουμε έτσι παθιασμένες συζητήσεις. Όσον αφορά όμως αυτό το ζήτημα της επικάλυψης, αυτή η μαγική λέξη, ε, λέξη συγγνώμη, η οποία ε, εξαπολύεται κάθε τόσο σαν πύραυλος έτσι ώστε ε, με ένα θαυμαστό τρόπο να διαγράψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή προβληματισμό. Μα στη Γαλλία έχουμε έναν στρατό και όταν ε, ε, αποφασίζουμε να βάλουμε ένα, ε, τη, τη σημαία του ΝΑΤΟ ή τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα σημείο στο οποίο είμαστε παρόντες, αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα σε χώρες, στις χώρες που βρισκόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την σημαία. Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν δέχονται ας πούμε τη σημαία του ΝΑΤΟ αλλά δέχονται ωραιότατα τη σημαία Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου του κ. Βανόρντε. Ναι, μπορεί να είναι έτσι αν έτσι θέλετε να το βλέπετε, αλλά υπάρχουν χώρες ε, ε, για τις οποίες οπωσδήποτε θα υπάρξει βέτο από πλευράς κάποιων μελών του ΝΑΤΟ σε ενδεχόμενη περίπτωση ε, αποστολής. Ας πούμε, εάν ε, η επιχείρηση στη Λιβύη γινόταν ε, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ δεν νομίζω ότι θα είχαν συμφωνήσει ε, όλοι. Απ' την άλλη πλευρά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και κάποιες αποφάσεις που αφορούσαν την Άγκυρα δεν θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί από όλα τα μέλη του, του ΝΑΤΟ. Nous sommes bien d'accord. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ακράδαντα το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πάει παντού και επομένως ε, ε, προκύπτει το ερώτημα ποιος θα πάει στις χώρες αυτές ε, και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση όσον αφορά την γεωπολιτική κατάσταση και θέση της. Ο κύριος Λίζεκ και μετά η κυρία Κοπά τελευταία για να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Μία επικοδομητική πρόταση. Είχαμε χιλιάδες συζητήσει πέρυσι από think tanks, από ιδρύματα για τη σχέση μεταξύ των στρατιωτικών δομών των ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας και το καθεξής. Μετά από τη συζήτηση αυτή φάνηκε ότι δεν είχαμε αρκετέ συζητήσει στο Κοινοβούλιο. Ίσως δεν έχουμε χρόνο, γιατί όλο ε, πρέπει να περάσουμε σε, σε την επόμενη έκθεση. Γιατί λοιπόν να μην διοργανώσουμε μια ξεχωριστή ακρόαση ή συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό φάνηκε από τη σημερινή συζήτηση. Και να προσκαλέσουμε και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Γιατί φαίνεται ότι μεταξύ μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το θέμα αυτό. the name of those guys? Ναι, ποιος ήταν ο Λούντιξ ο οποίος ε, έσπαγε τις ε, μηχανές. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνουν και οι πολιτικοί, λέει ο κύριος Πάσκου. Λοιπόν, η κυρία Κοπά, τελικά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ζωηρή, σφοδρή συζήτηση. Ήταν απαραίτητη εν ώψη και των ευρωεκλογών και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κυρίου Λίσεκ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε τη συζήτηση και στην Επιτροπή ε, και να μην περιοριστούμε μόνο σε τεχνικά ζητήματα, να εξετάσουμε και τη γενική εικόνα, γιατί μερικές φορές ε, χανόμαστε στις λεπτομέρειες και το εκλογικό σώμα θα πρέπει να καταλάβει καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Βανόρντεν, το θέμα των ε, Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι θέλουν να αποχωρήσουν, να ενδιαφέρονται περισσότερο οι Αμερικανοί πια για τον Ειρηνικό. Το, μάλιστα το στα τέλη του χρόνου, το τελευταίο τεθωρακισμένο των Αμερικανών θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Θα, οι μάχημες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα με μια ελαστική προσέγγιση να κάνουν κάτι όπου αυτό χρειαστεί. Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Ως προς τις επικαλύψεις, φυσικά συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. Ε, ζητούμε για την ε, αποφυγή της επικάλυψης, την ευθεία άμυνα, την ε, συγκέντρωση και συνεκμετάλλευση των πόρων. Όλα αυτά τα λέμε, αλλά είναι λόγια. Θα πρέπει να περάσουμε στα έργα. Όχι να λέμε απλώς ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δυνάμεις, να εξηγήσουμε και να βάλουμε με συγκεκριμένους όρους ε, τις απαιτήσει μα. Τι θέλουμε. Φυσικά δεν θέλουμε επικάλυψη, αλλά τι επιδιώκουμε. Δυστυχώ και πάλι εκτό μικροφώνου το σχόλιο του κ. Βαν Όρντεν. Oh, please, please, Mr. Van Orden, have, have a Now, uh, Mr. Campbell. Κύριε Κάμπελ, ε, μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνα είναι κάτι γνωστό τη φάση. Δεν θα το συζητήσουμε. Είναι διάταξη της συνθήκης. Οφείλουμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη, τελεία και παύλα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Θέλουμε την Μεγάλη Βρετανία στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως ε, ε, να αναχαιτίζει ή να τροχοπεδεί το όραμά μα το ρόλο μας ε, και τη σκέψη μα για το ρόλο που θέλουμε να παίξουμε στον κόσμο. Αυτό είναι ένα τίμημα που θα πληρώσετε κι εσείς και εμείς, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, συμφωνώ με τον Ανατονζό ότι η Αταλάντη στόχο έχει να προστατεύσει οποιοδήποτε πλοίο, φυσικά και τα πετρελαιοφόρα, τα δεξαμενόπλια και πρόσφατα πολλά δεξαμενόπλια τα κατέλαβαν οι πειρατέ. Έχουμε θέμα ενεργειακής ασφάλειας. Γιατί να αισθανόμαστε ε, ένοχοι. Από τη στιγμή που η ενεργειακή μας ασφάλεια υπονομεύεται από την πειρατεία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι σαφές. Θέμα προϋπολογισμού. Γνωρίζετε το θέμα του προϋπολογισμού είναι πολύ ευαίσθητο και λεπτό. Και στην δική μου πολιτική μου οικογένεια και στους Πρασίνου, γίνεται ολόκληρη συζήτηση γιατί λέμε ότι λυπούμαστε για την περικοπή των δαπανών, των στρατητικών δαπανών. Είμαστε κατά των δαπανών που ε, καταργούν ικανότητες που χρειαζόμαστε για να προσπίσουμε τους πολίτες, να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Είναι ένα πακέτο και τμήμα και της επικοινωνιακής μας στρατηγικής. Θα πρέπει να προβάλλουμε και σωστά επικοινωνιακά την ε, άμυνα. Γιατί μερικέ φορέ αισθανόμαστε ενοχέ όταν συζητούμε την άμυνα και το προσπαθούμε να το παρακάμψουμε. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Μα ενδιαφέρει η άμυνα. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να μεταφέρουμε καλύτερα επικοινωνιακά το μήνυμά μας στο κοινό. Φυσικά η Κύπρος είναι θέμα κλειδί για τη σχέση ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι να λυθεί το Κυπριακό δεν περιμένουμε ε, τα δύο, ε, τους να συνεργάζονται ομαλά και να συντονίζονται απρόσκοπτα. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος και στο θέμα αυτό. Κυρία Λέζινγκ, όταν μίλησε για ιδεολογία δεν ήταν προσβολή. Είναι διαφορετική προοπτική, αν θέλετε σε ό,τι αφορά το ρόλο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή απόψεων, να βρούμε ε, κοινά σημεία όπου υπάρχουν και να διαφωνήσουμε εκεί που έχουμε διάσταση. Αλλά μην το εκλαμβάνετε αρνητικά ή προσβλητικά. Έφυγε η κυρία Κρόνμπεργκ. Σίγουρα η Frontex δεν είναι αποστολή επιχείρηση της ΚΕΠΑ, αλλά είναι καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να σημαίνει προστασία εξωτερικών συνόρων. Αυτά και σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένω τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας και ε, η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Θέλουμε κοινή ευρωπαϊκή θέση και όχι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Είμαι πρόθυμη για συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή, η οποία βεβαίως θα συνεχιστεί, γιατί υπενθυμίζω ότι η 24 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, 24 ε, Σεπτεμβρίου ε, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα έχουμε μια δεύτερη συζήτηση την 14η Οκτωβρίου. Επομένως, ακονίστε τα επιχειρήματά σας για την 14 Οκτωβρίου και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί η έκθεση στην ΑΦΕΤ την 17η Οκτωβρίου έτσι ώστε να περάσει στην Ολομέλεια του ε, μηνός Νοεμβρίου. Περνάμε τώρα στη δεύτερη ε, έκθεση η οποία βεβαίως συνδέεται και με αυτήν που μόλις είδαμε, είναι η έκθεση του Μίκαελ Γκάλερ σχετικά με την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, ε, για την οποία έκθεση θα έχουμε την, ε, τις ίδιες προθεσμίες. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία ε, εκπονείται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ήτρε βάσει του άρθρου 50 και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα γνωμοδοτήσει επί του ιδίου θέματος, η ΙΜΚΟ. Ε, βασιστήκαμε και στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και άλλωστε είχαμε εδώ και ανταλλάξαμε απόψεις δύο φορές με τους Επιτρόπους Μπαρνιέ και Ταγιάννη. Πρόκειται για θέματα λοιπόν τα οποία έχουν ξανασυζητηθεί. Θα δώσω το λόγο στον Μίκαελ Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποτελεί σύμπτωση ότι ήρθε τώρα η ομάδα των επισκεπτών που έχω προσκαλέσει. Δεν τους ε, έφερα επίτηδες εδώ αυτή την ώρα για να με υποστηρίξουν. Και λοιπόν αυτή η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση της Άμυνας της Ευρώπης αποτελεί μια συμβολή ή τουλάχιστον μια απόπειρα συμβολής επικειμένη στις διασκέψεις κορυφής του Δεκεμβρίου, συμβολής λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πρωτίστως τους συντάκτες της φιλόδοξης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Πιεροντί και Καλπέλς από άλλη συναρμόδια επιτροπή. Συνεργαστήκαμε πραγματικά πολύ αποτελεσματικά με ε, τους δύο αυτούς συναδέλφους. Με ικανοποιεί και η από 24η έκτου ανακοίνωση της Επιτροπής και διαβεβαιώνω τους εκπροσώπους της εφόσον είναι παρόντες εδώ, ότι θα κάνω προσπάθεια οι προτάσεις τους όντως να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Για το σχέδιο εκθέσεώς μου, για την αφετηρία ορισμένα τα είπαμε ήδη, κρίσεις στην άμεση γειτονία μας, το μήνυμα των ΗΠΑ, καθίστε να ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι μόνοι σας Ευρωπαίοι με την σας, με τις γειτονικές σας περιφέρειες, το γεγονός επίσης ότι Έχουμε ασυντόνιστες περικοπές των αμυντικών προϋπολογισμών λίγο πολύ σε όλες τις χώρες μέλη και επίσης ασυντόνιστες αναδιαρθρώσεις των στρατιωτικών δομών των χωρών μελών. Απειλή απώλειας της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας βάσης μεταξύ άλλων διότι διάφορες επιχειρήσεις μετεγκαθίσταται σε τρίτες χώρες. Αν δείτε μάλιστα και τις πρόσφατες αναδιαθρώσεις της EADS, αλλά και τι είπε και ο ίδιος ο επικεφαλής της, είπε ότι στέλνουμε τους μηχανικούς μας εκεί όπου χρειάζονται και από τη στιγμή που φύγανε, φύγανε. Αν φύγουν δηλαδή από τον χώρο της στρατιωτικής βιομηχανίας και πάνε στον χώρο της πολιτικής, μη στρατιωτικής βιομηχανίας, τότε χάθηκαν πλέον για την βιομηχανία αυτή, η οποία άλλωστε επεκτείνεται και σε άλλες επεκτηνόμενες αγορές. Αυτή είναι η κατάσταση στην ε, Ευρώπη. Ιδρύθηκε ήδη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας από το 2004, που ήταν μια πρώτη απάντηση. Αυτός ο οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοδοτικά προβλήματα. Βεβαίως δεν είναι οργανισμός που φροντίζει για τις προμήθειες, είναι σαφές αυτό. Αλλά αναλαμβάνει και άλλα καθήκοντα και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να είναι μηδενικές οι αυξήσεις του προϋπολογισμού του. Ήδη από το 2007 έχουμε ανακοίνωση της Κομισιόν που καταστρώνει μια στρατηγική για μια πιο ενισχυμένη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Έχουμε και τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας που ήδη αυτά εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Άμυνας από το 2007. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουν κατατεθεί άλλες εκθέσεις υλοποίηση των υπεσχημένων και εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να επικριθεί. Έχουμε και το πακέτο για την άμυνα. Ακόμα δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα, ούτε υλοποιηθεί. Εν προκειμένου έχω να ασκήσω κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έννοια ότι δεν έχει πραγματική βούληση εφαρμογής του άρθρου 346 που επιτρέπει κατεξαίρεση στις χώρες μέλη εφόσον υπάρχουν πιεστικά εθνικά συμφέροντα να εξέρχονται της ενιαίας αγοράς. Κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για παντίους σκοπούς αλλά Αντιβαίνει όμως το πνεύμα της συνθήκης. Οι τρεις βασικές ιδέες του σχεδίου εκθέσεως έχουν ως εξή. Πρώτα, να δημιουργηθεί μια επιχειρησιακή, λειτουργική πολιτική που χρειάζεται βεβαίως μια στέρεα βιομηχανική βάση που να επιτρέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων για την εκπλήρωση των αποστολών. Δεν μπορούμε πολιτικά δηλαδή να αναλαμβάνουμε κάποιες δεσμεύσεις τις οποίες να μην μπορούμε μετά να υλοποιήσουμε στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να κάνουν έξτρα προσπάθεια και από την πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς και ότι η μετεγκατάσταση της βιομηχανικής μας βάσης σε τρίτες χώρες πρέπει να παρεμποδιστεί. Με το σχέδιο εκθέσεως προσπαθώ να δώσω ευρωπαϊκές απαντήσεις στα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι έχουμε, τι διαθέτουμε. Ποιες ικανότητες διαθέτουν οι χώρες μέλη. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε με ένα είδος ευρωπαϊκής απογραφής, μιας European Defense Review. Μακάρι αυτό να αποφασιστεί στην ε, διάσκεψη κορυφής. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για ασφάλεια και άμυνα για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές φιλοδοξίες με την δικαιολογημένη άλλωστε ζήτηση ε, στρατιωτικών ικανοτήτων. Για να υπάρξει πραγματικά μια διαδικασία ανάπτυξης ευρωπαϊκών ικανοτήτων χρειάζεται να ληφθούν τα ακόλουθα βήματα. Αφενός η εναρμόνιση των προμηθειών. Εναρμόνιση και συγχρονισμός προμηθειών και ε, ζητήσεως μάλλον και προμηθειών. Επίσης στην εκπαίδευση, χρήση και βελτίωση χρήσης των συστημάτων με στόχο την διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών μας δυνάμεων ήδη από την φάση των προμηθειών. Δεν έχει νόημα ο καθένας ασυντόνιστα να προβαίνει σε προμήθειες και μετά να εκπλήσεται ότι τα πράγματα αυτά δεν ταιριάζουν, δεν λειτουργούν τα μεν με τα δε. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα σφάλματα του παρελθόντος. Για παράδειγμα, το ελικόπτερο Τίγρης ή το μεταγωγικό αεροσκάφος 400 της ΕΡΒΑΣ που δεν έχουν ανταποκριθεί στις ε, απαιτήσει. Και πάρα πολλά παραδείγματα που έχουμε ποικίλε εκδόσεις εντό εισαγωγικών του ίδιου υλικού που όταν πάνε να χρησιμοποιηθούν από κοινού σε μια αποστολή δεν ταιριάζουν. Δεν έχει νόημα να γίνονται τέτοιε δαπάνε, τόσο μεγάλε δαπάνε, για να υπάρχουν τόσε πολλέ διαφορετικέ εκδόσει ενό τύπου υλικού. Εκτό αυτού, πρέπει να προωθηθεί η ευρωπαϊκή τυποποίηση και πιστοποίηση. Πρώτα, διαμεθοριακά, να διευκολύνουμε την πιστοποίηση και την, και την μακροπρόθεσμη ε, σύνταξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Security of supply, ασφάλεια προμηθειών. Αυτό είναι ένα κέριο θέμα που θα εξαρτηθεί από τις ικανότητες βιομηχανικής παραγωγής. Εδώ κυρίως ενδιαφέρει πού βρίσκεται η βιομηχανία αλλά δεν μας εξυπηρετεί να γίνεται η παραγωγή σε τρίτες χώρες. Τώρα για την αδιασφάλιση των προμηθειών. Ρωτώ, γιατί δεν μπορούν οι χώρες μέλη να υποσχεθούν οι μεν στις δε ότι θα δίνουν για τις εξαγωγές γενικές ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τις εξαγωγές. Αυτό θα βελτιώσει την δυνατότητα εξαγωγών. Αυτό μπορεί να συζητηθεί και μέσα στην μόνιμη διαρθρωμένη ανταλλαγή απόψεων. Αυτό που να γίνει και μέσα στην ομάδα ευρώ ή μεταξύ των χωρών Σένγκεν και ούτω καθεξής. Έχουμε δηλαδή τις βάσεις για να προωθήσουμε την ιστορία αυτή. Τώρα, η διάθεση βασικών τεχνολογιών, key enabling technologies, είναι σημαντικό να συντονιστούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΟΑ. Χρειαζόμαστε δηλαδή στρατηγική των δύο αυτών φορέων που να εξασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε τεχνολογίες κρίσιμες για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Τέλος, έρευνα και ανάπτυξη. Το οφείλουμε στον συνάδελφό μας Έλερ ότι περιλήφθηκε η μη στρατιωτική έρευνα για τον ορίζοντα 2020 πρέπει να συνδυαστεί με τη στρατιωτική έρευνα και χαίρομαι για την πρόταση της Κομισιόν για προπαρασκευαστικά μέτρα για την αμυντική έρευνα. Σημαντικό είναι να ενταχθούν τα μέτρα αυτά γρήγορα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε και σύμφωνα με το άρθρο 185 της συνθήκης να καλυφθεί χρηματοδοτικά το πλαίσιο αυτό μέχρι ότου ισχύσει το επόμενο πλέον χρηματοδοτικό πλαίσιο. Όταν το 2009 Συμβούλιο και Κοινοβούλιο εξέδωσαν το λεγόμενο πακέτο της άμυνας, παρόλες τις εθνικές επιφυλάξεις στο άρθρο 346 που είναι δυνατόν βέβαια να υποβληθούν αλλά πρέπει να είναι αιτιολογημένες, αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι οι εθνικοί οργανισμοί προμηθειών να θέτουν κατά κανόνα, να κάνουν κατά κανόνα τις ε, προσκλήσεις ε, εκδήλωση ενδιαφέροντος πανευρωπαϊκά. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς δεν πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση μέσω του υπερβάλλοντος ύλου της ε, αμυντικής γραφειοκρατίας ορισμένων χωρών. Θετικό παράδειγμα για μένα είναι η Σουηδία, η οποία όταν επιθυμεί να κάνει μια προμήθεια για τις αμυντικές της δυνάμεις εξετάζει πρώτα εάν μπορεί να προμηθευτεί το σχετικό υλικό από την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά για την εκθεσή μου και αναμένω τις παρεμβάσεις, είτε επικοδομητικές είτε άλλες. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στο, στο σκιώδη συγγητές, πρώτα στον κύριο Ζέμκε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας και να ξεκινήσω από την θετική ε, κρίση για το σχέδιο αυτό του κύριου Γκάλερ Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη η υποβολή αυτής της έκθεσης. Είναι κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα της ε, κοινή ε, βιομηχανικής ε, και τεχνολογικής βάσης της άμυνας. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί αρχίζει και γίνεται γνωστό και να ευαισθητοποιείται περισσότερο και η πολιτική ότι αυτό το θέμα είναι θετικό και θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Τεχνολογική ε, Βάση Άμυνας. Αυτό είναι το θετικό σχόλιο. Υπάρχουν όμως και τρία προβλήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί η επίλυση αυτών των τριών προβλημάτων κατά τη γνώμη μου θα επηρεάσει ε, θετικά το έγγραφο ώστε να γίνει και καλό αλλά και να έχει και μεγάλη ε, πιθανότητα να πραγματοποιηθεί, να μεταφερθεί στην πράξη. Και το θέμα δεν είναι να πούμε μερικά ωραία πράγματα, αλλά να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Να δώσουμε σε αυτό το έγγραφο σάρκα και ωστά Θα επισημάνω λοιπόν μερικά προβλήματα για να αθαρρύνω μερικά κρατημέρη να ε, υποστηρίξουν την θέση μας. Το πρώτο θέμα. Βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε λίγο πολύ Έξι χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία, να συγκεντρώνουν το 80% του, του αμυντικού δυναμικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Οι αποφάσεις μας θα ενισχύσουν ε, το ρόλο των επιχειρήσεων αυτών των χωρών ή θα δημιουργήσουμε όρους ε, και συνθήκες ώστε και άλλες χώρες οι υπόλοιπε 22 χώρε, γιατί παραλαμβάνω μιλούμε για 6 χώρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28. Ή θα μπορέσουν λοιπόν με τι προτάσει αυτέ και άλλε χώρε να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τουλάχιστον μερικά τμήματα τη αμυντική του βιομηχανία. Εγώ θα ήθελα η ανάπτυξη αμυντική βιομηχανια να γίνει σχετικά ισορροπημένα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και Πολωνία έχει θετική γνώμη για τα αντισταθμιστικά ωφέλη, ενώ άλλε χώρε έχουν διαφορετική γνώμη, η Πολωνία είναι υπέρ του offset. Γιατί θεωρούμε ότι ε, είναι καλό τρόπο για μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Δεύτερο ζήτημα. Χρειάζεται πραγματικά να συζητήσουμε αυτό το Συμβούλιο για τον αμυντικό κλάδο ή θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε απλώς το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο πολλαπλασιασμός των οργάνων δεν εξασφαλίζει η λύση των προβλημάτων. Ίσως καλύτερος τρόπος θα ήταν να ενισχύσουμε το ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, που ούτως ή άλλως έχει συγκεντρώσει κάποια πείρα και ε, θα μπορέσει να να επιλύσει τα προβλήματα. Προτιμώ αυτή τη θέση λοιπόν να ενισχύσουμε τη θέση της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Τρίτο τώρα θέμα, όταν ε, μιλούμε για το δυναμικό, το εξοπλιστικό, το αμυντικό μας, θα πρέπει να απαντήσουμε και στην ερώτηση τι, ποιο είναι το οικονομικό αντικείμενο του, της αμυντικής βιομηχανίας. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε το αντικείμενο του οικονομικού κλάδου της αμυντικής βιομηχανίας. Αν γίνει αυτός ο ορισμός μπορούμε εύκολα να λύσουμε και το πρόβλημα της ε, ολοκλήρωσης της ένταξης του. Ε, ε, δεχτήκαμε με τον Κρυσίστο Φιλίσεκ ε, αρνητικές ειδήσεις. Χθες η Ολλανδία ε, αποφάσισε για 35 Eurofighter παρόμοιες, παρόμοια σχέδια έχουν και οι Ιταλοί και άλλες χώρες. Αυτές οι επιλογές δείχνουν ότι αν δεν τονίσουμε την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης όχι μόνο δεν θα αναπτυχθεί περαιτέρω αλλά θα εξαφανιστεί γιατί φαίνεται ότι πολλές χώρες προτιμούν τις αμερικανικές προμήθειες. Ευχαριστώ πολύ Νταφ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλωσορίζω την έκθεση αυτή του κυρίου Γκάλερ που παίζει σημαντικό ε, ρόλο στην ε, συνολική προσέγγιση την οποία να προσπαθούμε να επιτύχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά ζητήματα άμυνας και ε, ασφάλειας. Νομίζω ότι σωστό είναι να κατακρίνουμε τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, τα οποία ε, ε, δίνουν όλο και περισσότερες δίνουν όλο και περισσότερο βάρος στους ώμους της αμυντικής βιομηχανίας χωρίς όμως να αλλάξουν τις συνθήκες ελπίζω ότι στην επόμενη επικαιροποίηση της ε, συνθήκης ε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις όσον αφορά την ΕΟΑ και φαντάζομαι ότι και η Κομισιόν θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο και από πιο κοντά με το θέμα. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να πούμε κάτι εδώ για την Τουρκία. Μιλήσαμε προηγουμένως για το ζήτημα της ε, Κύπρου σε σχέση με το ΝΑΤΟ στα πλαίσια της έκθεσης ε, ε, ΚΟΠΑ. Υπάρχει όμως και ένα σημείο αδυναμίας στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε ε, και την Τουρκία σε αυτό το εγχείρημα. Τι μπορεί να πει ο κύριος Γκάλερ όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ. Εμείς είμαστε από αυτούς που βλέπουν θετικά την έκθεση και συμφωνούμε απολύτως ότι ε, το πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, ε, κάνουν μια πολιτική εξαγωγών η οποία τελικά αποβαίνει επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει συσχετισμός ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα εδώ είναι να βρεθούν λύσεις, ε, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορεί να υπερκεραστεί ο κατακαιρματισμός, ε, πώς μπορούν να καλυφθούν ε, τα, οι ελλείψεις της αξιοπιστίας ή της εμπιστοσύνης, πώς μπορούν να αποφευθούν οι επικαλύψεις. Ε, οι οδηγίες ε, για, τις, ε, για την ασφάλεια και για την άμυνα είναι, πηγαίνουν προς τον καλό δρόμο όσον αφορά τώρα του τον Εθνικό Οργανισμό Προμηθειών κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι οι πληροφορίες σωστές αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξουν μαζικές αγορές εξοπλισμού, κυρίως όσον αφορά οχήματα στρατιωτικά. Θα πρέπει να γίνει κάτι λοιπόν. Επίσης ε, για τις ε, προμήθειες ε, ακούμε ότι η Ρουμανία θέλει να αγοράσει παλιά ε, πολεμικά αεροσκάφη χωρίς όμως ε, να κάνει ε, συγκεκριμένη διαδικασία πρόσφυσης ενδιαφέροντος πράγμα που σημαίνει ότι η Eurofighter και κάποια άλλη ευρωπαϊκή ή σουηδική εταιρεία δεν μπορεί να συμμετάσχει. Όσον αφορά το, τα χρήματα, ίσως αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. δεν ε, λέμε ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα να ε, συμπεριλάβουν και την άμυνα. Ε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Πάσκο ότι υπάρχουν τροποποιήσεις πλέον και ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός και οι περισσότερες χώρες δυσκολεύονται αλλά νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά επιστημονικά προγράμματα δεν θα πρέπει να κατευθούν με την άμυνα. Το ίδιο ε, ισχύει και για, την, ε, ε, για τον οργανισμό άμυνας. Δεν πρέπει να στηρίζεται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει τα ίδια τα κράτη να κάνουν, να στηρίξουν τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν ε, ίδιους ε, πόρους, ε, ίσως και με τη βοήθεια, με κάποια εξωτερική βοήθεια, αλλά πάντως τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεργαστούν και όσον αφορά την έρευνα και όσον αφορά ε, την, τον ΕΟΕ. Καλωσορίζουμε και την έκθεση και τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούζινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη συζητήσαμε προηγουμένως αρκετά θεμελιώδη θέματα. Τώρα εδώ θα έρθω σε ορισμένες λίγες επικοδομητικές παρατηρήσεις. Γράφετε στην έκθεσή σας, κύριε Γκάλερ, στο σχέδιο εκθέσεώς σας διαπιστώνεται ότι για να αντιμετωπιστεί η εγχώρια ζήτηση πρέπει να εξάγουν, για να, μάλλον για να αντισταθμίσουν την εγχώρια ζήτηση που μειώνεται εννοείται, να εξάγουν περισσότερο σε τρίτες χώρες. Το θεωρείται αυτό αναγκαιότητα για την ε, αμυντική βιομηχανία, για την εξοπλιστική βιομηχανία δεν θεωρείτε ότι η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια ενίσχυση του ελέγχου των εξαγωγών εξοπλισμών. Αυτό δεν το βλέπω στην έκθεσή σας. Γιατί δεν ζητήσατε να συνταχθεί και τέτοια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μου φαινόταν εμένα πολύ σημαντική. Και να περιληφθεί η διάσταση αυτή δηλαδή στην έκθεσή σας. Ευχαρίστως να σας συνδράμω στην ε, προσπάθεια αυτή. Κύριε Κάλερ, επίσης έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Κρόνμπερκ. Στο άρθρο 4 της εκθέσεώς σας γράφεται ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας η βιομηχανία και η διαστημική βιομηχανία έχουν λάβει τώρα μία έξτρα διάσταση. Ακριβώς σε αυτό που αναφέρθηκε η κυρία Κρόνμπερκ προηγουμένως την διάδραση μεταξύ ε, ε, αμυντικής και μια ε, στρατιωτικής βιομηχανίας. Μιλάτε εδώ εμέσως για χρηματοδότηση, διότι το 40 παράγραφος 2 της συνθήκης λέει ότι η χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται αμυντικών δηλαδή και άλλων τέτοιων διαστάσεων δεν επιτρέπεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αναφέρεται αυτό άραγε και στη χρηματοδότηση της αμυντικής έρευνας. Συμφωνείτε με την ερμηνεία αυτή ή θεωρείτε ότι δεν είναι σωστή. Και θα ήθελα να ακούσω άλλωστε και την άποψη άλλων συναδέλφων. Ο κύριος Τέρχο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τον εισηγητή για το σχέδιο εκθεσής του. Πιστεύω ότι το σχέδιο αυτό αποτελεί μια καλή βάση και δεν έχω να προσθέσω και πολλά γιατί το θέμα αυτό μπορεί να μην είναι της μόδας αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν η Ευρώπη θέλει μια αξιόπιστη άμυνα αν θέλει να έχει επιχειρησιακή ικανότητα και να γίνει σημαντικός παράγοντας είτε σε περιφερειακό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, αν θέλουμε να είμαστε χώρος τεχνολογικής ανάπτυξης θα πρέπει να υλοποιήσουμε τους στόχους του εγγράφου. Δεν θα υποβάλω καν τροπολογίες να φανταστείτε. Ευχαριστώ κύριε Κοπά. Thank you very much, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μάικλ Γκάλερ για την έκθεσή του γιατί είναι ακριβώς αυτό που θα πρέπει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Γενική Συζήτηση. Γνωρίζουμε ότι εν μέσω της πιο σοβαρής οικονομικής κρίσης από το 30 δεν έχουμε περισσότερα κονδύλια για την άμυνα. Θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στους πολίτες πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής Τεχνολογική βαϊσάμινα γιατί και θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ε, καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Τα περισσότερα προϊόντα που παράγονται στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία έχουν διπλή χρήση, στρατιωτική και πολιτική. Και το θέμα της διπλής χρήσης ακριβώς δημιουργεί πρόβλημα στην δημιουργία ορθωτικών γραμμών, όπως είπε η κυρία Κρόνμπερκ. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε λοιπόν την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε ισχυρότερε ενέργειε μεταξύ τη έρευνα και στο στρατιωτικό και στον πολιτικό τομέα, ώστε να έχουμε καινοτομία με λιγότερη επιβάρηση του προπολογισμού. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία ανάμεσα στην στρατιωτική και μη έρευνα ε, ε, για μας σαν πολιτική ομάδα ε, θα πρέπει η οποιαδήποτε τροποποίηση στην βιομηχανία αυτή να συνοδεύεται από μέτρα τέτοια τα οποία θα μετριάσουν το κοινωνικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι ε, ε, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία σε αυτές τους χαλεπούς καιρούς του στην περίοδο κρίσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη βιομηχανία, θα πρέπει να στηρίξουμε και την καινοτομία και την έρευνα ε, και μέσω αυτής της μεθοδολογίας θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να προχωρήσουμε μπροστά προσωπικά εγώ αλλά και ως εισηγήτρια για το προηγούμενο θέμα κοινή πολιτική Είμαι απολύτως ευτυχής με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και μάλιστα θα προσπαθήσω να συζητήσω με τον Μάικλ Γκάλερ για να δούμε εάν ε, μπορούμε να προωθήσουμε κάποια κοινά στοιχεία ε, των δύο εκθέσεών μας. Αλλά ε, και τελειώνω με αυτό, θα πρέπει να βρούμε κάποια κεντρικά σημεία τα οποία θα προωθήσουμε για να περάσουμε σαφή μηνύματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκου. Σας ευχαριστώ. θα ήθελα να πω ότι πέραν του γεγονότος ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι η αξία και το πλεονέκτημα της έκθεσης είναι ότι είναι συνοπτική. Και με στή. Εστιάζει την προσοχή μας και τη σκέψη μας στα πιο κέρια ζητήματα. Και Όλα αυτά που αναφέρει η έκθεση είναι ακριβώς αυτά τα σημαντικά πεδία. Γι' αυτό είμαι υπέρ της έκθεσης. Γιατί φαίνεται ο κόσμος ε, έρχεται και πληρώνει ένα διαγώνα, αλλά φαίνεται σαν είναι στημένος. Γιατί βλέπετε ότι για πολλέ εκθέσει συμπίπτουν οι απόψει του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών και των άλλων ομάδων. Αυτό όμω δεν οφείλεται στο γεγονό ότι πλησιάζουμε προ τι ευρωεκλογέ, αλλά ότι πλησιάζουμε προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνες. Και έχουμε πολλές προσδοκίες από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υποστηρίζω την έκθεση λοιπόν και συγχαίρω τον εισηγητή τη. Ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει πάλι ο εισηγητή μα. Μην ξεχνάτε ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι ίδια... Είναι ίδια με την προηγούμενη έκθεση, 24 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη συζήτηση θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, ίδιες προθεσμίες με την προηγούμενη έκθεση. Ο Μάικλ. Ευχαριστώ. Θα ακολουθήσω τη διαδική σειρά των παρεμβάσεων. Κύριε Σέμκε, μιλήσατε για ορισμένα πράγματα. Είπατε ότι οι μεγάλες χώρες, όλες μαζί, οι μεγάλες χώρες, έχουν το 80% του αμυντικού προϋπολογισμού και να δώσουν την ευκαιρία και σε άλλες χώρες μικρότερες. Ναι, σαφώς ναι. Σε πολλές χώρες Υπάρχει γνώση και ικανότητα των βιομηχανιών τους δηλαδή, ανεξαρτήτως του γεγονότος από το αν κάθε μια από αυτές τις βιομηχανίες είναι και ανταγωνιστική, ανεξάρτητα από αυτό. Νομίζω αυτό πρέπει να εξετάσουμε είναι να μην έλθουμε σε μια κατάσταση όπου αυτό το άρθρο 346 να ενεργοποιείται από ορισμένε χώρε μόνο και μόνο επειδή έχει σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο ένα ειδικό εργοστάσιο το οποίο θέλει ντε και καλά να το διατηρήσει στη ζωή για κάποιο διάστημα ακόμα. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλα εργαλεία έτσι ώστε από τη μια μεριά να δούμε από τα διαρθρωτικά ταμεία για παράδειγμα πώς μπορεί να προκύψει μια διαρθρωτική προσαρμογή σε διάφορες περιφέρειες έτσι ώστε να διατηρηθούν και κάποιες θέσεις απασχόλησης στον τεχνολογικό τομέα. Αυτό ίσως είναι ένας τρόπος να δούμε όπου υπάρχει δηλαδή υπερβάλλουσα ικανότητα να μπορέσει να μειωθεί. Και αυτό όχι μόνο στις μικρές χώρες, μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Για παράδειγμα σε μεγάλες χώρες έχουμε σαφώς υπερβάλλουσα ικανότητα, πλεονάζουσα ικανότητα. Άρα λοιπόν διαρθρωτικές αλλαγές να τις έχουμε πάντοτε ως ενδεχόμενο υπόψη μα για να αποφύγουμε ενδεχόμενα προβλήματα. Πάντως οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τη συνεργασία ώστε η ικανότητα και η γνώση να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν εποφελώς από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται. Ακριβώς μετά από την διάσκεψη κορυφής για την άμυνα χρειαζόμαστε και ένα επίσημο συμβούλιο το οποίο να φροντίσει να βρει τρόπους υλοποίησης των όσων θα συμφωνηθούν μεταξύ άλλων. Αυτή δηλαδή η τεχνητή ας πούμε παραλλαγή που έχουμε, δηλαδή ανεπίσημα συμβούλια Υπουργών Άμυνα ή από κοινού με του Υπουργού Εξωτερικών. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, αλλά για τα όσα προέλθουν από το συγκεκριμένο αυτό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητηθούν επισήμω πλέον σε Συμβούλια Υπουργών Αμήνη. Βεβαίω, να ενισχυθεί και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα αλλά και το Συμβούλιο της ε, άμυνας. Για την ερώτηση του κυρίου Νταφ για την ε, προσαρμογή των θέσεων, του της θέσεως μάλλον του ΕΟΑ με τις θέσεις της Κομισιόν. Εγώ έχω κάνει και την πρόταση το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας να πληρώνεται από τον προϋπολογισμό της Κομισιόν. Αυτό για μένα αποτελεί μια δυνατότητα. Προ την κατεύθυνση αυτή. Τώρα αν θα πούμε κάτι εδώ σχετικά με την Τουρκία. Εάν κατορθώσουμε ο ΕΟΑ και ο ΟΚΑΡ να συγχωνευτούν, σκέλος του ΝΑΤΟ δηλαδή, να μπορέσουν να συγχωνευτούν επαναλαμβάνω, πριν να συμμετάσχει στον ΟΚΑΡ η η Τουρκία, η οποία θέλει να μπει και στον Ευρωπαϊκό, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, είπα ότι εγώ φοβούμαι ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μπορεί η Τουρκία να προβάλλει κάποιο βέτο. Να δούμε τώρα εάν ΕΟΑ και ο ΟΚΑ μπορούν να συνεργαστούν με κάποιο τρόπο και τότε ευχαρίστως να μπει και η Τουρκία. Αλλά να είναι μέσα η Ένωση ως Ένωση και επομένως να μην μπορεί πλέον η Τουρκία να προβάλλει βέτο. Για την κυρία Κρόνμπεργκ, Ορίζον 2020 και αμυντική έρευνα, η στρατιωτική πολιτική έρευνα, όπως είπε η κυρία Κοπά, όλα αυτά είναι σχεδόν διτής χρήσεως στον τομέα αυτό, dual use. Για μένα είναι άλλωστε συμφωνημένη πολιτική στον τομέα της άμυνας επιτρέπεται να υποστηρίζει, το λέει αυτό και η συνθήκη, επιτρέπεται να υποστηρίζεται και με πόρους της έρευνας. Στη συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι μπορούν να υποστηρίζονται χρηματοδοτικά από τους πόρους μας και άλλοι τομείς συνεργασίας της Ένωσης. Και μάλιστα εφόσον είναι, αν συμφωνεί και ομόφωνα, διοντολογικά υποστηρίζονται. Δεν είναι χειρότερη οι τομείς αυτοί από άλλους. Και για το εξωτερικό εμπόριο της Ένωσης Εάν στείλουμε τώρα το αυτοκίνητο, νοσοκομιακό αυτοκίνητο ή φτιάξουμε το σχολείο ή στείλουμε το θωρακισμένο όχημα, για μένα αυτά τα πράγματα είναι το ίδιο αιτιολογημένα, το ίδιο θεμελιωμένα στις πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι ηθικά απορριπταία. Γι' αυτό εντάσσονται στις πολιτικές της Ένωσης και άρα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της έρευνας. Σε ό,τι αφορά τον τομέα ελέγχων, εξαγωγών, εξοπλισμών, εάν ενισχύσουμε τη δική μας βάση, αν φεύγει κάτι από εμά να εξαχθεί προς τα έξω, τότε έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε καλύτερα τις συμφωνίες για τους ελέγχους εξοπλισμών. Να μην φτάσουν δηλαδή εξοπλισμοί σε λάθος χέρια. Αν όμως εμείς δεν κάνουμε τίποτα εδώ και οι εταιρείε παραγωγής εξοπλισμού σηκωθούν και φύγουν και πάνε και μετεκατασταθούν σε τρίτες χώρες, τότε δεν έχουμε απολύτως κανένα έλεγχο πλέον του τι εξάγουν. Τα πλαίσια υπάρχουν. Τα πλαίσια, το πλαίσιο ειδικά για τους ελέγχους είναι σωστό, είναι ορθό. Μπορώ να το περιλάβω βεβαίως ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Αλλά νέους κανόνες δεν νομίζω να χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ άλλωστε την κυρία Κοπά και τον κύριο Πάσκου και τον κύριο Ζέμ και βεβαίως των σοσιαλιστών για την υποστήριξη που προσφέρουν στο σχέδιο εκθέσεων. Ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ξανά έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την έκθεση. Πάντως, για να επανέλθω σε ένα από τα θέματα που έθιξε ο Μάικλ, η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και, και το γεγονό ε, το κατά πόσο θα επιφορτήσει ένα Συμβούλιο Υπουργών μετά, ε, Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, να ξεπεράσει αυτές τις τακτικές ε, συνεδριάσεις και να αναλάβει συγκεκριμένες εξουσίες και ένα συγκεκριμένο δικό χάρτη για θέματα για τα οποία θα μπορούν να λάβουν αποφάσεις ε, αυτό θα ήταν ε, αν όχι θεαματικό αρκετά σημαντική πρόοδος γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε μία ακόμη άτυπη συνάντηση υπουργών άμυνας ωραίες ε, συμπαθητικές ε, αυτές οι συναντήσεις αλλά από θεσμική άποψη δεν έχουν και μεγάλη αξία. Και καλό θα ήταν και για τη βιομηχανική και για την επιχειρησιακή πτυχή τα Συμβούλια Υπουργών Άμυνας ε, να έχουν πιο επίσημο χαρακτήρα και δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Το απόγευμα θα έχουμε μία συνεδρίαση για το ΣΕΣΑΡ και την εφαρμογή του συστήματος ε, ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού για, στρατιωτική, για το στρατιωτικό τομέα. Και φυσικά έχουμε και εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις. Πολλές και διάφορες. Σας ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη.